Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα στη μέση διάταξη πρέπει να τα συζητήσουμε. Το σημείο 2 λοιπόν είναι η εξέταση της έκθεσης ε, ε, συλλογής στοιχείων στη Λάρνακα και η παρουσ... και... το, το θέμα και το σημείο 40 επίσης δεν το έχουμε έτοιμο στην τελική του εκδοχή για σήμερα. Σας παρακαλώ να σημειώσετε ότι η συνεδρίασή μας το απόγευμα θα ξεκινήσει στις 3.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΦΚΟ PHS P1α002 και μας προσκαλεί η ΑΦΚΟ ω συνδεδεμένη επιτροπή με βάση το άρθρο 55 για μια παρουσίαση από τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμαντ τη νέα πρόταση για κανονισμό για την πρωτοβουλία των πολιτών. Πολύ σημαντικό να ε, είναι παρούσα και η επιτροπή μα. Θα πάμε εκεί για μια ώρα και στις 4.30 ε, θα συνεχιστεί σε αυτή την αίθουσα η τακτική μας συνεδρίαση και θα πρέπει να ξεκινήσει η συνεδρίαση τάχιστα. Μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε έτσι την ημερήσια διάταξη και να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης του Οκτωβρίου. Τα έχετε δει. Ωραία, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις της Προέδρου. Διάφορα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε απευθείας στη μελέτη ο ρόλος ε, της Επιτροπής Αναφορών στα πλαίσια της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που την παρήγγειλε το Τμήμα Πολιτικής ΣΥ μετά από δικό μας αίτημα. Και είναι πολύ κατάλληλη και η στιγμή για να τη συζητήσουμε και θα απολαύσουμε και ένα PowerPoint. Ο κύριος Μάρκ Πρίσλι, που είναι καθηγητής για θέματα πολιτικής αναπηρίας και επιστημονικός ε, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, Εμπειρογνωμόνων για άτομα με αναπηρία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μας ξανακαλέσατε φέτος. Ε, είναι η συνέχεια της μελέτης που είχε ζητήσει η ΠΕΤΗ καταρχήν το 2015. Μια πιο πλατιά μελέτη για την ανάλυση των αναφορών και μελέτη η οποία είχε επικυρωποιηθεί το 2016. Τώρα καταγράφουμε τις φετινές ε, εξελίξεις και ορισμένες προκλήσεις για το μέλλον. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι το 1 τέταρτο περίπου του εκλογικού σώματος στην Ευρώπη δηλώνει ότι έχει κάποιου βαθμού αναπηρία ή ε, αισθητηριακή στέρηση. Και αυτοί ψηφίζουν. Ίσως είναι η μεγαλύτερη μειοψηφία του εκλογικού σώματος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται επίση ε, στο κέντρο τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προσιλωμένο στην προάσπισή του και στην δημιουργία μια Ευρώπη των δικαιωμάτων. Επίση, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε αναγνωρίζονται όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά και στο διεθνέ δίκαιο. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ε, ε, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει συνάψει στο στο ίδιο επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Ε, είναι το μόνο μέρος αυτής της ε, σύμβασης που δεν είναι κράτος. Η μελέτη μας ε, βρίσκεται στο site της ΠΕΤΗ, στο ίντερνετ. Είναι μια πολυσέλιδη σελίδα, αξιολογεί το πλαίσιο στο οποίο κινείται η σύμβαση του ΟΗΕ πλαίσιο της, ε, του προστατευτικού ρόλου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των αναπήρων και την ανάλυση των αναφορών που έχουμε λάβει τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια στις οποίες αναφέρονται θέματα αναπηρίας. Δεν πρόκειται να σας πω πάρα πολλές λεπτομέρειες γι' αυτό. Το σημαντικό είναι να δούμε πού εντάσσεται η ΠΕΤΗ μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ποιος είναι ο ρόλος της ΠΕΤΗ σε σχέση με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Ο ρόλο αυτός έχει σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, ένα, έχει μια υποχρέωση με βάση τη Σύμβαση να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την προστασία, την παρακολούθηση και την ε, προώθηση των δικαιωμάτων. Και η ΠΕΤ είναι θεματοφύλακα, ιδιαίτερα όταν κάτι δεν πάει καλά. Όμω, ε, όχι μόνο στην προστασία, αλλά και στην προώθηση των δικαιωμάτων έχει ρόλο η ΠΕΤΗ και στην ε, υποβολή κάποιων εκθέσεων ε, τακτικά για την κατάσταση των δικαιωμάτων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχική έκθεση συμπεριλάμβανε μια σειρά συστάσεων. Ε, θα τις ε, βρείτε στο τέλος των ε, σημειώσεων που σας, του ενημερωτικού σημειώματος που σας υπέβαλα. για να συνοψίσω, έχουμε έναν αριθμό μηχανισμών εντός των ευρωπαϊκών οργάνων, μηχανισμών προστασίας. Δεν είναι μόνο η πέτη τμήμα αυτού του συνόλου. Ε, έχουμε την διαδικασία αναφορών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε και μια διαδικασία ε, προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή. Έχουμε μια αντίστοιχη διαδικασία ε, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας και τέταρτον υπάρχει ένας μηχανισμός υποβολής παραπώνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε η ΠΕΤΗ εντάσσεται σε ένα πανόραμα διαφορετικών μηχανισμών που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες πολύ συγκεκριμένες και πολύ σημαντικές όμως αναφορές φτάνουν στην Επιτροπή ΠΕΤΗ και αυτό ε, καθιστά την ΠΕΤΗ ιδιαίτερα σημαντική. Τα συμπεράσματα της προηγούμενης μελέτης ήταν ότι, όπως είπαμε, οι ε, ανάπηροι, τα άτομα με αναπηρίες είναι σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού ε, και μάλιστα ψηφίζουν περισσότερο κατά μέσο όρο και περισσότερη ποσοστία από ότι ε, τα άτομα που δεν έχουν αναπηρίες. Το βασικό πόρισμα της ανάλυσης των αναφορών είναι ότι ε, μη ε, δικαστικές απαντήσεις δεν λύνουν πάντοτε τα προβλήματα των αναφερόντων πολλές από αυτές τις αναφορές δεν οδηγούν σε λύση των προβλημάτων του αναφερόμενου. Οπότε η Επιτροπή προσπαθεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει άλλες διαδικασίες, να πιέσει εκεί που μπορεί, ε, εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται τις αρμοδιότητες με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Και όταν δούμε τις φετινές αναφορές αυτό επιβεβαιώνεται. Πολλές αναφορές, ε, αναφορές σχετίζονται με την κοινωνική προστασία, την απασχόληση, την προσβασιμότητα εντός των κρατών μελών που έχουν σχέση με, κατά κάποιο τρόπο με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά που σε μεγάλο βαθμό αποτελούν ε, κοινέ αρμοδιότητες. Πρέπει να δούμε πώς η Επιτροπή ΠΕΤΗ επηρεάζει αυτή τη διαδικασία επιμερισμού των αρμοδιοτήτων και πώς επιτελεί συντονιστικό έργο. Ε, επικαιροποίηση 2017. Ε, ενημερωτικό σημείωμα. Ε, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων. Καταρχήν να δούμε τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ε, την σύμβαση του ΟΗΕ, υπέβαλε και μια δήλωση αρμοδιοτήτων ε, στον ΟΗΕ, όπου ανέφερε τις, ε, τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες για άτομα με αναπηρίες. Ήταν όμως μια, ένας κατάλογος ε, ενδεικτικός, όχι εξαντλητικός το 2016 επικαιροποιήθηκε επί τη βάση και ε, μελετών του ακαδημαϊκού δικτύου. Το σημαντικό είναι όμως ότι δεν υπάρχει ένας απλός τρόπος ε, να υποβάλουμε ε, ή να επεξεργαστούμε κάποιον εξαντλητικό κατάλογο αρμοδιοτήτων. Γιατί οι αναπηρίες θα πρέπει να ενταχθούν ως οριζόντιο θέμα στις ευρωπαϊκές πολιτικές όπως και το φύλλο. Οπότε αυτή η διαδικασία είναι ατέρμονη. Το mainstream λοιπόν της αναπηρίας, των αναπηριών είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Ε, για παράδειγμα, σε όλους αυτούς τους τομείς εδώ που αναφέρω. Δεν θα τους σχολιάσω όλους, αλλά θα δείτε για παράδειγμα το πώς έγινε αυτό πέρσι ε, στο Κοινοβούλιο, για παράδειγμα ε, με τη δημιουργία του ε, δικτύου CRPD. Έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα εργασίας 2017-2019 στο, στην διακοινοβουλευτική ομάδα. στο πώς οι αναπηρίες θα αντιμετωπίζονται στην περιοχή, στις υποένταξη χώρες. Ε, οι αναπηρίε ε, συμπεριλήφθησαν στην ετήσια έκθεση της ΠΕΤΙΑ του 2016, διοργανώθηκε και ένα εργαστήρι στις 12 Οκτωβρίου. Όλες αυτές είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι οι αναπηρίες αναγνωρίζονται κατά προτεραιότητα. αυτή είναι μια πρακτική την οποία θα πρέπει να επενέσουμε. Παρόλο ότι σε ορισμένες ε, περιπτώσεις το θέμα αυτό εξαφανίζεται σε ορισμένου τομεί, ας πούμε, ε, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έχει γίνει δουλειά σε αυτό. Ε, η ΠΕΤΗ ζήτησε μια ε, έκθεση για τις... διακρίσεις, καθώς επίσης και για την, το νόμο περί προσβασιμότητας. Είχαμε μια σημαντική αναφορά ε, για το θέμα αυτό πέρσι και νομίζω ότι η Πέτη το πρόθεσε πολύ ε, προσεκτικά. Και για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία είχαμε ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, οπότε ε, εισακούεται η φωνή της Πέτη στο Κοινοβούλιο. Επίσης βλέπουμε και κάποια παραδείγματα νομοθετικών εξελίξεων Το κεκτημένο είναι πολυπλατεία, αλλά έχουμε την ε, σύναψη της ε, συμφωνία του Μαρακές, ε, που ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη, την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προσβασιμότητα των κρατικών ε, sites στο ίντερνετ, την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Νόμου περί προσβασιμότητας, ε, ε, όπως ζήτησε ο δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά η ΠΕΤΗ ζήτησε την σύντομη υιοθέτηση αυτού του νόμου. Πέραν όμως της, των εξελίξεων, έχουμε και παραδείγματα στην, στον συντονισμό των πολιτικών. Οι αναπηρίες εξακολούθησαν να είναι ορατές σε διάφορα μέτρα συντονισμού, ίσως δεν είναι το, νούμερο ένα θέμα προτεραιότητας. Αλλά συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα της αποϊδρυματοποίησης στο συντονισμό των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιο σημαντικά όμως παραδείγματα που είδαμε είναι οι προσπάθειες της Κομισιόν να διασφαλιστεί ότι οι αναπηρίες θα αντιπροσωπευτούν στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στις ανοιχτές μεθόδους. Εκεί είναι μια σημαντική ευκαιρία για όλους μας να ενθαρρύνουμε την Κομισιόν ε, να εντάξει ε, την προοπτική αυτή σε όλες τις διαδικασίες που είναι δυνατόν. Πολλές από τις αναφορές που έφτασαν εδώ έχουν σχέση άμεσα με την κατάσταση σε ένα κράτος μέλος το οποίο ε, βρίσκεται ε, στο μεγεθυντικό φακό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σε τέτοιου είδους λοιπόν ε, περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται σημασία και στις αναπηρίες. Ε, στην, στην, στα θεμελιώδη δικαιώματα επίσης γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε οι ε, αναπηρίες να παραμείνουν ε, μέσα στο ραντάρ ε, και τα 19 θέματα έτσι και αλλιώς έχουν σχέση με κάποιο τρόπο <clears throat> με την αναπηρία, οπότε θα πρέπει και εκεί σε όλα αυτά τα ζητήματα να ενταχθεί και η αναπηρία. Επίσης βλέπουμε πρόοδο και στο Eurostat για το θέμα των δεδομένων το σχετικό με τις αναπηρίες το, η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των σχετικών με τις αναπηρίες και της ανισότητας μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία και δεν έχουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία στις βασικές ευρωπαϊκές έρευνες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση στην επισκόπηση την, ε, για το εργατικό δυναμικό. Οπότε δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αριθμούς, ε, τον αριθμό, να υπολογίσουμε τον, ούτε καν τον αριθμό των ε, εργαζόμενων αναπήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε όμως θετικές εξελίξεις. Ε, η, υποομάδα των δικτών της Επιτροπής Σοσιοκοινωνικής Προστασίας επεξεργάζεται δείκτες κοινωνικής προστασίας που λαμβάνουν υπόψη την αναπηρία η εισαγωγή των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον, στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ ε, απαιτεί την ανάλυση των ε, στοιχείων της αναπηρίας σε, σχέση με τους 19 στόχους, οπότε και αυτό είναι πολύ θετικό. Και τέλος, κοιτούμε τις αναφορές που ήρθαν φέτος εδώ στην ΠΕΤΗ, το είδαμε και στο αστείο του Οκτωβρίου, βλέπουμε ποια θέματα υπογραμμίζονται είναι τα ίδια ακριβώς με αυτά των προηγούμενων εκθέσεών μας. Για παράδειγμα προσβασιμότητα, αλλά και σε σχέση με άλλα θέματα απασχόλησης κοινωνικής προστασίας κλπ. Um, so the remaining... Λοιπόν, ας δούμε τώρα και τις υπόλοιπες διαφάνειες. Αναφέρομαι εδώ πέρα στις κοινέ προκλήσεις που προκύπτουν από το πλαίσιο το οποίο σας περιέγραψα η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όταν αναφέρθηκε στην πρόοδο που είχε σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε στην ευθύνη που φέρει να ενσωματώσει τη διάσταση αναπηρία σα σε βασικέ πολιτικέ όπω η απασχόληση, η εκπαίδευση και άλλοι τομεί κοινωνική πολιτική. Και νομίζω πραγματικά ότι έχουμε εδώ πέρα μια χρυσή ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Είχαμε βέβαια και κάποιε εξελίξει στον συντονισμό του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύμβαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ζητήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, έκανε συγκεκριμένε προτάσεις προκειμένου το πλαίσιο αυτό να παραμείνει ανεξάρτητο, αυτόνομο και να υπάρχουν συγκεκριμένοι πλέον μηχανισμοί συντονισμού. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε κάποιες σημαντικές προκλήσεις, σημαντικές ευκαιρίες καταρχάς μας δίνονται τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει μια επανευθυγράμμιση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Άνομα με Αναπηρίε με την εφαρμογή τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου από το 2016 τη κυρία Χέλγα Στίβεν, κάλεσε και αυτή για μια σφαιρική αναθεώρηση τη στρατηγική για την αναπηρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα αναπηρίε από το 2021 στο 2030 και περιμένουμε τώρα να δούμε πώ θα εξελιχθεί στο μέλλον η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική για την περίοδο, όπω σα είπα, 2021-2030. Το χρονοδιάγραμμα όμω πολιτική είναι κρίσιμη σημασία σε σχέση με τι προκλήσει και τι ευκαιρίε που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η περίοδος αυτή, η μεταβατική προς μια νέα στρατηγική, η ευθυγράμμιση στρατηγικής αυτής με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει νέες προτάσεις, νέες εκθέσεις μάλλον πρόοδου προς τα Ηνωμένα Έθνη σε σχέση με τη στρατηγική αναπηρία. Και ουσιαστικά Συνάδει αυτό και με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα έχουμε βέβαια και μία νέα επιτροπή, ένα νέο κοινοβούλιο σύντομα. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή ευθυγράμμισης της νέας στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες με όλες τις υπόλοιπες σημαντικές πολιτικές και τις σημαντικές εξελίξεις που θα δούμε στο μέλλον στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα βέβαια έχουμε το θεματολόγιο των ΗΕ του 2030 το οποίο συνάδει με το χρονοδιάγραμμα για τη νέα στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες και η νέα αυτή λοιπόν στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονιστεί με το θεματολόγιο των ΗΕ το 2030. Θεωρώ πάντω ότι έχουμε πολύ σημαντικέ ευκαιρίε προκειμένου να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική που θα συνάδει με το θεματολόγιο των ΗΕ το 2030. Και καλείται βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο τη Σύμβαση των ΗΕ. Αυτό το έχει ζητήσει και η δική σα επιτροπή αλλά και άλλοι σημαντικοί παράγοντε. Έχουμε βέβαια σημαντικές ακόμα προκλήσεις μπροστά μας, να καταφέρουμε δηλαδή να εξισορροπήσουμε το πλήρε και σφαιρικό πεδίο εφαρμογή τη σύμβαση CRPD των ΗΕ με το πιο περιορισμένο εύρο των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε πώ επιτροπές αντιδικήσεις στην Επιτροπή Αναφορών, θα τοποθετηθούν σε αυτή τη συζήτηση, πώ θα καταφέρετε να επηρεάσετε και να προστατεύσετε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίε σε αποκλειστικέ αρμοδιότητε και σε συντρέχουσε αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να δούμε επίση ποια θα είναι η δομή, η εντολή και η σύνθεση του νέου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύμβαση CRPD, ιδίως στα πλαίσια του νέου προαιρετικού πρωτοκόλου. Όπως και σε προηγούμενες εκθέσεις αναφερόμαστε στις αρχές των Παρισίων, θεωρούμε ότι ε, θα πρέπει αυτές να κατευθύνουν τη διαμόρφωση οποιοδήποτε νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης έχουμε και τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου λέγεται εκεί πέρα ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και όπου λέγεται εκεί πέρα ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση όσον αφορά μια ανάληψη κοινή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και σε ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Εμεί σα ευχαριστούμε και πολλέ φορέ στην ε, Επιτροπή μα ε, έχουμε την εντύπωση ότι κατακλυζόμαστε από πάρα πολλέ αναφορέ για το ζήτημα αυτό. Στα πλαίσια όμω τη τρέχουσα θητεία, νομίζω ότι καταφέραμε πολλά σημαντικά πράγματα, άρα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μα. Κάνουμε πολλά πράγματα και καταφέραμε σημαντικά επιτεύγματα, τίποτα δεν έχει κλείσει, τίποτα δεν είναι τέλειο ακόμα, αλλά νομίζω ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη. Ιδιαίτερα περήφανη. κύριε Πρίστλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωσή σα αυτή σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη που κάνατε. Είχατε έρθει και πέρυσι, είστε εδώ και φέτο και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, θα έλεγα για μας, να μπορούμε να έχουμε το συνεχιζόμενο αυτό διάλογο μαζί σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ σήμερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η κυρία Μακουλάδα Παλένθια Πορέρο έχει το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθήσαμε την πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η Επιτροπή σας με πολύ ενδιαφέρον γιατί κάνει μια πολύ καλή επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στην πολιτική για τις αναπηρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμεριζόμεθα σε πολλά σημεία τις απόψεις του καθηγητού Πρίστλη και εργαζόμεθα για να βελτιωθεί η κατάσταση και να αντιμετωπιστούν τα κενά που διαπιστώθηκαν. Θα αναφερθούμε σε ορισμένα σημεία. Πρώτον, για το ενωσιακό πλαίσιο. Πριν από δύο μήνες, για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι το σημείο επαφή στα πλαίσια της σύμβασης συναντήθηκε με το νοσιακό πλαίσιο και εκπονεί ε, τις μεθόδους συνεργασίας και εντοπίζει διάφορες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Ο καθένας από την δική του πολύ διαφορετική οπτική γωνία. Τα μέλη του πλαισίου το οποίο είναι πλαίσιο και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ως πλαίσιο έχει ε, γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο. Έχει υιοθετηθεί από το Συμβούλιο. Η χρηματοδότηση των διαφόρων φορέων ε, γίνεται αυτόνομα, αλλά να τονίσω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, έχουν γίνει διάφορες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ε, είμαστε στη φάση εντοπισμού των ευρωπαϊκών μη ομικρών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν είτε επισήμως στο πλαίσιο είτε απλώς να συμβάλλουν στην επιτήρηση της εφαρμογής της ε, σύμβασης. Τώρα για τα στατιστικά στοιχεία και την ε, επιτήρηση. Πρώτον, μπορούμε όλο και περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε στατιστικά στοιχεία για ε, την παρακολούθηση των ε, δικτών για διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής και ε, οι στόχοι STG περιέχουν διάφορους δείκτες για, την, ε, για τις αναπηρίες. Σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε ε, θα συζητήσουμε τους ε, κοινωνικούς δείκτες τους, ε, συγγνώμη, τους δείκτες της αναπηρίας για, στα πλαίσια του πλαισίου για την κοινωνική πολιτική. Ελπίζω να υπάρξει θετική κατάληξη και έτσι θα γίνει πιο ε, επίσημη η διαδικασία συλλογή στοιχείων στα πλαίσια δικτών για τα άτομα με αναπηρία. Βέβαια πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν υπάρχει ένας αποφασισμένο, ένας ε, επίσημος δείκτη για την σύνδεση μεταξύ απασχόλησης και αναπηρίας. Κάνουμε κάποιες εξομοιώσεις για να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία ε, από πλευράς απασχόλησης. Αλλά θα θέλαμε να εντάξουμε κάτι τέτοιο στις μελέτες που κάνουμε για το εργατικό δυναμικό. Για τη στρατηγική, ο κύριος Πρίσλι ε, αναφέρθηκε σε ορισμένα αποτελέσματα. Και φυσικά τονίζουμε ότι οι στόχοι της κύριας έκθεσης της Κομισιόν εξακολουθούν να ισχύουν. Πρέπει να συνεχιστεί η εργασία για να επιτύχουμε όλα τα αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο θα δούμε αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε σε δύο χρόνια. Υπήρξε μια περίοδος συζήτησης όπου κάναμε διαβουλεύσεις και με άτομα με αναπηρία και, και τους οργανισμούς που τους εκπροσωπούν αλλά θέλουμε να υπάρξει και μία ανεξάρτητη αξιολόγηση για τα αποτελέσματα της στρατηγικής μας πριν αρχίσουμε να εκπονούμε το νέο πλαίσιο πολιτικής για τις αναπηρίες που ακόμη πρέπει να καθοριστεί. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που θέσατε αυτό το θέμα στην πρώτη γραμμή και κάνετε μια καλή επισκόπηση της διαδικασίας ε, εν μέσω της οποίας ε, βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Και τώρα συνάδελφοι, ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πρίστλεϊ για την ε, μελέτη την οποία έκανε και την έκθεση που μας ε, παρουσίασε και να επισημάνω δύο-τρία θέματα. Πρώτον, το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών. Διότι αυτές ε, οι δεκάδες, εκατοντάδες ε, παρεμβάσεις, αναφορές που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια από άτομα με ειδικέ ανάγκες και ο ρόλος της Επιτροπής, ο οποίος είναι σημαντικός, ανέδειξε πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως την Επιτροπή Αναφορών ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Δεύτερον, δημιούργησε ένα βήμα παρέμβασης ε, και ε, προτάσεων εκ μέρους των ίδιων των ατόμων με ειδικές ανάγκες που μας εξηγούσαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Μάλιστα την προηγούμενη, στην προηγούμενη συνεδρίασή μας είδαμε πώς υποφέρουν άτομα με ειδικές ανάγκες στη Ρουμανία που δεν έχουν πρόσβαση στους ε, ρουμανικούς ε, σιδηροδρόμους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο νομίζω πρέπει να το καταγράψουμε στα θετικά της δραστηριότητας της Επιτροπής Αναφορών και φυσικά ως ένα μηχανισμό σύνδεσης των πολιτών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι οι υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ε, σύμβασης του ΟΗΕ ε, για την προστασία των ατόμων ε, με αναπηρία, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δρά εν κενό, δεν υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, υπάρχουν υποχρεώσεις όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οφείλει στο πεδίο αρμοδιοτήτων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ε, σύμβαση του ΟΗΕ. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο και νομίζω ότι απλά το ότι στέλνει ένα κείμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ποιες αρμοδιότητες έχει δεν νομίζω ότι δίνει απάντηση. Θα πρέπει να δει με ποιες πολιτικές πρωτοβουλίες θα συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις που έχει ε, από την Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των ατόμων με ειδικέ ε, ανάγκες. Το τρίτο θέμα είναι πρακτικά ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την έκθεση της συναδέλφου, της κυρία Στίβενς που ανήκει και στο ECR, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία όλων των θεμάτων για να μπορούμε πραγματικά ε, να έχουμε ένα ουσιαστικό ρόλο. Και τέλος, θα έλεγα ότι το ζήτημα της στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι ένα θέμα πρώτα απ' όλα ηθικό. Είναι θέμα υποχρέωσης της ίδιας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των, ε, πολιτών, και των Ευρωβουλευτών για τη στήριξη αυτών των ατόμων. Επομένως, ακόμη και αν δεν ήταν μεγάλος ο αριθμός, δυστυχώς είναι μεγάλος αριθμός, αλλά ακόμη και αν είχαμε ελάχιστους ε, συμπολίτε μας, ε, με, άτομα με ειδικές ανάγκες, πάλι τα ίδια έπρεπε να κάνουμε. Δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα χώρο όπου υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν και οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και άρα εμείς έχουμε ένα κοινό μια constituency στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε, Ακόμη και ένας να ήταν και δέκα να ήταν θα έπρεπε να έχουμε κάνει τα ίδια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πρώτο βήμα σημαντικό να δούμε παρακάτω κυρία Πρόεδρε τι άλλες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρουμε για να στηρίξουμε τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. now I would like to Ευχαριστώ. Η Ρώσα Έστερας. Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ τον ομιλητή για τη μελέτη που μας παρουσίασε. και εγώ έχω διάφορες ερωτήσεις και προς την Μακουλάδα από την Κομισιόν. Οι αναφορές μας μπορούν να παίξουν ρόλο καταλήτη για να εντοπίσουμε τις αδυναμίες των κρατών μελών στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Με ανησυχούν διάφορα και με απασχολούν. Πρώτον, δεν αναφέρεται αρκετά ο διαχωρισμός αναφύλων τα ειδικά προβλήματα των γυναικών δηλαδή, στις μελέτες για τα άτομα με αναπηρία. Όλες οι στρατηγικές, είτε για τα θέματα της αναπηρίας, είτε για τα θέματα ισότητας των φύλων, δεν λαμβάνουν υπόψη ειδικά το θέμα των γυναικών με αναπηρίες. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αυτών των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ε, σεξουαλική ζωή, στη ζωή της γενικότερα, σε όλους τους τομείς. και επανειλημμένα. Το έχουν απαιτήσει και τα Ηνωμένα Έθνη επανειλημμένα. Πρέπει όλα τα θέματα και όλες οι μελέτες να λαμβάνουν υπόψη και να ε, μετράνε συγκεκριμένα τα προβλήματα των γυναικών με αναπηρίες. Να ξέρουμε τι χρειάζονται. Βεβαίω η συνθήκη του Μαρακέ ήταν ε, σημαντική και σημαντική ήταν ε, και η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητα. Ξεκίνησε ο τριμερής διάλογος, αλλά η Κομισιόν έχει ζητήσει μία πράγματα που είναι ανεπαρκή μεν, αλλά περισσότερα από όσα υπήρχαν. Και ε, βεβαίως ξέρουμε ότι δεν θα είναι πάντα προσβάσιμες όλες οι υπηρεσίες και όλες οι μορφές ε, μεταφορικών μέσων γιατί οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν φυσικά να αναλάβουν το κόστος άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δική μας Επιτροπή μέσω του τριμερούς ε, διαλόγου να εμείνουμε στη στάση της Επιτροπής γιατί φοβάμαι ότι το Συμβούλιο με βάση τη γενική του πρακτική περικοπών βεβαίως στις διακηρύξεις όλοι συμφωνούν αλλά μετά, όταν πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, λένε υπάρχει οικονομικό κόστος και πάντα οι νόμοι αυτοί έχουν μεταβατικές περιόδους για να γίνουν οι αναγκαίες βελτιώσεις και αυτές οι μεταβατικές ε, διατάξεις τελικά διαιωνίζονται. Αυτό βλέπουμε και με, ε, με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη που νομίζω ότι έχει καθυστερήσει. Πρέπει να τονίσουμε ότι η θέση μας είναι πραγματικά υπέρ της εφαρμογής της σύμβασης αυτής. Και τώρα, μετά ο κοινωνικός πυλώνας. Υπεγράφει πριν από δύο εβδομάδες στο Γκέτεμπουργκ και τώρα είναι πραγματικά η κόρη του οφθαλμού μας. Αλλά το θέμα είναι και να εφαρμοστεί γιατί αναφέρεται η εκπαίδευση που να τους συμπεριλαμβάνει όλους, ισότητα ευκαιριών, αξιοπρεπής εργασία, ανεξαρτησία, όλα τα θέματα που αναφέρονται και στην έκθεσή μας. Αλλά ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Θα παραμείνουν λόγια. Και νομίζω ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν μπουχτίσει πολύ ωραίες διακήρυξεις, λίγα στην πράξη. Βεβαίω, καθυστερεί η Ευρώπη. Καθυστερεί η λήψη αποφάσεων. Για να αποφασίσουμε κάτι χρειάζονται τρία χρόνια. Οπότε τουλάχιστον η Επιτροπή μας θα πρέπει να αγωνιστεί με την μακουλάδα στην Κομισιόν και με όλους που μπορούν να μας βοηθήσουν για να είμαστε η φωνή των ατόμων με αναπηρία. Γιατί ξέρω ότι αυτός ο Ευρωπαϊκός Χάρτης πήγε στην Ήτρε και υπήρξαν καταστροφικές επιπτώσεις. Γιατί πάντα το οικονομικό υπερισχύει του κοινωνικού. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και από την Πρόεδρο που ξέρω πόσο αποφασιστικά βοηθάει να γίνει η Επιτροπή μας σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της ε, σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ Ρόζα. Ξέρω ότι είναι κάτι με το οποίο πραγματικά σας συναρπάζει, αλλά σας παρακαλώ να μακρηγορείτε γιατί δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο. Και τώρα η κυρία Καμπεθόν Ρουίθ. Να ευχαριστήσω και τον ε, ε, υπεύθυνο της ε, έκθεσης, πολύ σημαντική και λεπτομερής. Θα ήθελα και εγώ να σημειώσω το ρόλο της Επιτροπής μας γιατί νομίζω πως είμαστε μία από τις επιτροπές ε, που ε, πραγματικά είναι προσιλωμένη στην βοήθεια των ατόμων με αναπήρεια. Δεν ξέρω αν θα χρειαζόταν μια ειδική επιτροπή, όπως λέει η έκθεση, στο Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι ε, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και αυτή την πρόταση. όπως είπε η Ρόζα Σταράς, ε, μερικές φορές ε, οι αναπηρίες μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο. Η σύμβαση του Μαρακές και άλλα θέματα τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικά και δείχνει ότι είμαστε προσιλωμένοι προς αυτό το στόχο. Ε, δεν θα πω τίποτα άλλο για τον κοινωνικό πυλώνα, όπως είπε η Ρώσα, αλλά θέλω να επιμείνω στο θέμα του φίλου. Είναι κάτι το οποίο επανέρχεται διαρκώς. Ε, πόσο δύσκολο είναι να ε, υιοθετήσουμε δείκτες που να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την αναπηρία αλλά και το φίλο μέσα στην αναπηρία. Να αναλύσουμε δηλαδή τα στοιχεία αναφύλλο. Εγώ θα συμπεριλάμβανα και δύο πρόσθετους δείκτες. Με, με ανησυχούν ιδιαίτερα τα παιδιά και τα άτομα με, νοητική αναπηρία. Γιατί έχουν ένα θέμα προσβασιμότητας πιο ε, οξύ από τους υπόλοιπους. Θα ήθελα να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε μηχανισμούς για τον εντοπισμό και την καταγραφή των παιδιών και των ατόμων με νοητική αναπηρία, διανοητική αναπηρία. Αν δούμε τις αναφορές που φτάνουν, αφορούν άτομα με σωματικές αναπηρίες, όχι με διανοητικές τόσο πολύ πνευματικές αναπηρίες. Θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και να αγγίξουμε και αυτούς και τα παιδιά και να συμπεριλάβουμε αυτές τις δύο ομάδες ως δείκτες στις επόμενες εκθέσεις μας. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Soledad. Beatriz Becerra. Θα είμαι σύντομη, δεν θα επαναλάβω επιχειρήματα άλλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πρίστιλ για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να επισημάνω ότι συμφωνώ 100% με τα επιχειρήματα και τις ανησυχίες της Ρώσα Εσταράς. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες για το φύλλο, είναι απόλυτος απαραίτητοι. Είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε αποτελεσματικοί στο οριζόντιο συστηματικό έργο που πρέπει να κάνουμε. και το θέμα της ε, προσβασιμότητας πρέπει να ειδωθεί από αυτό το πρίσμα. Και τρίτον, κοινωνικός πυλώνας. Θα πρέπει οι συμφωνίες, οι μεγάλες συμφωνίες να υποστηρίζονται με κονδύλια. Γιατί αλλιώς ε, μένουμε στα λόγια. Η ομάδα των φιλελευθέρων υποστηρίζει την εφαρμογή της σύμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των θεμελιών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες. Τα δικαιώματα τα δικά τους και των οικογένειών τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έχει καταγραφεί και στα, σε ευρωπαϊκές συμφωνίες και στις διεθνείς συμφωνίες. Θέλουμε όλα τα κράτη-μέλη να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ. Υποστηρίζουμε την ε, διεύρυνση της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, EU Disability Card. Θέλουμε να διευκολυνθούν τα άτομα με αναπηρίες ε, στην μετακίνησή τους, στις μετακινήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς να υπογραφεί η συνθήκη του Μαρακές ε, με την ανάληψη όλων των ευθυνών που σημαίνει αυτό. Ε, καλωσορίζουμε την ε, νομοθεσία για την πρόσβαση στα, σε κρατικά site στο ίντερνετ και στην προσαρμογή των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχει νομίζω έχουμε μια σειρά κοινών στόχων, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ευχαριστώ λόγω στην κυρία Ντανόκα και μετά θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το θέμα. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Ένα ερώτημα το οποίο θέλω να, θέσω, να θέσω σε σχέση με την κάρτα αναπηρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μπεθέρα το έθεσε αυτό πριν από λίγο. Δεν κατάλαβα πάντως πολύ καλά τις παρατηρήσεις που κάνατε όσον αφορά την αφορά 1500 του 2016 όπου είπατε ότι μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα παρόλα αυτά αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας Μήπως θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο για το ζήτημα αυτό όσον αφορά το ζήτημα της αρμοδιότητας και τις δυνατότητες ε, χρησιμοποίησης, εισαγωγής μάλλον της κάρτας αυτής και αν μη τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε μία μελέτη για να δούμε τελικά πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε την απόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν δηλαδή ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν τέτοιες κάρτες αναπηρίας, αλλά πάλι όχι. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων με αναπηρίες και θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση. Σας ευχαριστούμε κυρία Στανόκα και ευχαριστούμε και εσάς κύριε Πρίσλεϊ. Για το συγκεκριμένο αυτό ερώτημα νομίζω ότι θα μπορούσατε διμερώς να το συζητήσετε και θα πρέπει να προχωρήσουμε και στα επόμενα σημεία της μερίστα διάταξης. Προτού πάμε στο επόμενο σημείο, θα ήθελα να σας πω ότι το 2020 είναι ο νέος κύκλος υποβολής εκθέσεων και αυτό είναι πραγματική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε τι έχουμε κάνει σε σχέση με τη συστάση του 2015 των ΗΕ, τι πρόοδο έχουμε σημειώσει και αν θα μπορούσαμε τελικά να ευθυγραμμίσουμε την πρόοδο αυτή με την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ και μπορείτε να έρθετε διμερώς σε επαφή με την κυρία Σντανόκα για να απαντήσετε στο ερώτημά σας. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε γρήγορα στο επόμενο σημείο της μερίστης διάταξης και θα ήθελα να καλωσορίσω τους αναφέροντες από την Φιλανδία. Φτάσατε, πολύ ωραία. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην αφορά 1394 της Πία Ματιχάλδη, εξ ονόματος του Ιδρύματος για τα άτομα με νοητική στέρηση, με πολλές υπογραφές αναφορά αυτή, σχετικά με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες προμήθειες και την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο που εισάγει διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Έχετε το λόγο για δυόμιση λεπτά ο καθένας. Αναφέρομαι στην κυρία Ματιχάλτη, στον κύριο Χίλτουνετ και στον κύριο Βίρκαμάκη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που δέχθηκε την αναφορά μας. Η κόρη μου η Γέννη ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη μονάδα ομαδικής στέγασης ε, Καγκρασού Ροσκού από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η μονάδα. Κάθε πέντε χρόνια ο πάροχος υπηρεσιών αλλάζει και την τελευταία φορά που έγινε αυτό, η εταιρεία η οποία ανέλαβε τις υπηρεσίες αυτές εκχώρησε τις υπηρεσίες αυτές μετά από δέκα μόνο μήνες. Ξέρετε ότι όλες αυτές οι αλλαγές προκαλούν τεράστια αναστάτωση στους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις μονάδες ομαδικής στέγασης και υπάρχει και ένα πρόβλημα με το προσωπικό, γιατί ξέρετε ότι οι νέοι αυτοί με αναπηρίες εξοικειώνονται με το προσωπικό, το οποίο μετά μετακινείται σε άλλες μονάδες. Και αυτό προκαλεί τεράστια σύγχυση και τεράστιο άγχος στην καθημερινή ζωή των νέων αυτών με αναπηρίες και βέβαια να στατώνει και τη ζωή και του ίδιου του προσωπικού πλαισίωσης και υποστήριξης. Φανταστείτε ότι είναι σαν να έχετε κάθε πέντε χρόνια ένα νέο σύντροφο, ο οποίος φτάνει στο σπίτι σας, ζει μαζί σας και σας λέει πώς θα πρέπει να ζείτε, πώς θα πρέπει να τρώτε, πώς θα πρέπει να χειρίζεστε τον ελεύθερο χρόνο σας. Αυτό προκαλεί τεράστια οδύνη και τεράστιο στρες σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις ε, μονάδες ομαδικής ε, στέγασης. Ξέρετε ότι ε, οι νέοι εκεί αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα, πολλές φορές καταλήγουν να διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα. Η κόρη μου Γέννη που ήταν μια πάρα πολύ εύθυμη πρόσχαρη κοπέλα Βλέπω τώρα ότι δεν θέλει καν να επιστρέψει σε αυτή τη μονάδα ομαδική στέγαση κάθε φορά που να μα δει, εμένα και τον πατέρα τη. Ξυπνάει ξαφνικά στο μέσο της νύχτας και ζητά να κοιμηθεί στο κρεβάτι των ε, γονιών της, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι 29 ετών άλλωστε. Και το πρόβλημα είναι ότι το προσωπικό δεν γνωρίζει καθόλου ποιες είναι οι καθημερινές ανάγκες της και ουσιαστικά παραμελούν κάποιες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες των καθημερινών αναγκών της ε, Γέννη. Ξέρετε ότι η Γέννη περπατούσε πάρα πολύ στο παρελθόν, έκανε πάρα πολλέ βόλτες Τώρα δεν τη δίνεται καν η ευκαιρία αυτή να βγει από αυτή την ομάδα, μονάδα ομαδική στέγασης. Όταν ζούσε μαζί μας έκανε πάρα πολλές τέτοιε βόλτες, πολλούς περιπάτους, ενώ τώρα διανύει μια ζωή πολύ πιο καθιστική και καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά την κάνει να οπισθοδρομεί. Η κατάστασή τη επιδεινώνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υπηρεσίε αυτές για τα άτομα με αναπηρία να είναι πιο σταθερές. Αν δεν είχαμε όλους αυτούς τους αλλεπάλους κύκλους εξωτερικής ανάθεσης, θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ πιο εύκολα. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος, ή μάλλον η κυρία Χίλτουνετ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Ο Άντι Αϊταλάσκο, ο γιος μου, είναι ένας νέος με ειδικέ ανάγκες ο οποίος στεγάστηκε αυτό σε μια μονάδα μοναδική στέγασης και χρειάζεται παρακολούθηση και υποστήριξη σε 24ωρη βάση. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ομιλίας, χρησιμοποιεί τη νοηματική, χρησιμοποιεί τα χέρια του, τα δάχτυλά του, και βέβαια η δυνατότητα επικοινωνία που έχει είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Χρησιμοποιεί μια περιορισμένη μορφή νοηματική γλώσσα και ελάχιστοι τελικά μπορούν να τον καταλάβουν και να επικοινωνήσουν μαζί του. Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουμε να τον καταλάβουμε καλύτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι θέλει να πει με τις κινήσει κινήσεις τις οποίες κάνει με τα χέρια του. Και το πρόβλημα είναι ότι όσο λιγότερο γίνεται κατανοητός, τόσα περισσότερο είναι τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν μεταξύ του άντι και του υπεύθυνου προσωπικού. Ξέρετε ότι α, τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι του ζητήθηκε να μπει σε συγκεκριμένα ιδρύματα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επίσης, η αλλαγή του προσωπικού στις μονάδες ομαδικής στέγασης, στις οποίες διαμένει, έχει προκαλέσει πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά προβλήματα. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλη αναστάτωση στον Άντι και έχουν ε, βέβαια μειώσει και την αυτοπεποίθησή του. Εξαιτία αυτή τη διαδικασία δημοσίων διαγωνισμών, το προσωπικό σε αυτέ τι μονάδε ομαδική στέγαση αλλάζει συνεχώ. Από ό,τι φάνηκε, κύριο μέλημα ήταν η μείωση του κόστου. Μα είπαν ότι θέλουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην πράξη όμω για τον Άντι τίποτα δεν γίνεται πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη πραγματικέ του ανάγκε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίρκαμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. Ο τρόπος με τον οποίο ε, οργανώνει η Φινλανδία μέσω πρόσκλησης ε, για εκδήλωση ενδιαφέροντος ε, της υπηρεσίας προς με αναπηρία παραβιάζουν τους κανόνες ε, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε χιλιάδες άτομα με αναπήρες στη Φιλανδία και όλα αυτά θίγουν και τα άτομα αυτά και τους ε, οικείους τους. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών είναι κατά λοιπόν αυτής της σύμβασης γιατί δεν δίνει καμία ε, δυνατότητα να επιλεγούν οι σωστοί πάροχοι υπηρεσιών. Έχουμε σαφείς ενδείξεις στη Φιλανδία ότι τα άτομα με αναπηρία και οι γονείς τους δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ε, ε, ενστάσεις και παράπονα για διοικητικές αποφάσεις που τους αφορούν. Κάτι που θα πρέπει να μπορεί να γίνει σε ένα κράτος δικαίου. Η μεγαλύτερη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η Φιλανδία δεν επιτρέπει να υπάρχει η σωστή σχέση μεταξύ των ε, φροντιστών και των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να επιτρέπεται να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ε, για να μπορούν να, να παρασχεθούν σωστά αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά με αυτές τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και την αλλαγή του παρόχου κάθε πέντε χρόνια γίνεται μια βίαιη αλλαγή ε, στη ζωή των ατόμων αυτών. Και έχουμε σαφείς αποδείξεις για το τι άγχος προκαλούν αυτές οι αλλαγές στα άτομα με αναπηρία. Τι πίεση και στρες. Η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες της Ένωσης έχει στόχο να διασφαλίζει τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτές τις διαδικασίες. Αλλά στη Φιλανδία παρατηρούμε τη δημιουργία ιδιωτικών μεγάλων μονοπωλίων για τις υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρίες είναι κάτι που ε, συμβαίνει και ευρύτερα στις υπηρεσίες υγείας. Οπότε κάνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μια συνέχεια στη βοήθεια που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία. Υπάρχει και η πρωτοβουλία των πολιτών όπου 72.000 πολίτες έχουν υπογράψει μία αναφορά αλλά η κυβέρνηση λέει ότι δεν ε, υπάρχει καμία δυνατότητα ανάληψης δράσης γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει ότι οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται μέσω της διαδικασίας καθορισμού παρόχων που προβλέπει η οδηγία. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσχέρειες και δεν το καταλαβαίνουν τα άτομα με αναπηρίες ούτε και οι γονείς τους. Έτσι ε, η νομιμοποίηση και η αποδοχή της Ένωσης ε, στα μάτια των φιλανδών πολιτών μειώνεται πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το σύστημα αυτό ε, για τις δημόσιες προμήθειες δεν χρησιμοποιείται σε ορισμένες άλλες χώρες. Και όπως και με τον Brexit δεν καταλαβαίνουν τα επιχειρήματα. Επιπλέον, έχουμε στείλει πολλές αναφορές και θα υποβληθεί και μία άλλη αναφορά που θα σας υποβάλουμε για την ε, προμήθεια διερμηνέων νοηματικής για άτομα με δυσχέρειες ακοής. Πρόκειται για ε, του διερμηνεί που ε, έδιναν βοήθεια σε χίλια άτομα και τα οποία ξαφνικά άλλαξαν. Οι οποίοι ξαφνικά άλλαξαν. Ο πρόεδρο, ε, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική στιγμή τη δραστηριότητά μα. Έχουμε απασχοληθεί με το θέμα αυτό. Αν ακούσετε τον καθηγητή προηγουμένω για να μας ενημερώσει ε, είναι σαφές ότι η Επιτροπή μας ε, αποδίδει μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά αλλά θα επανέλθουμε ας ακούσουμε την κυρία Λούπη που είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους αναφέροντες που μας ενημέρωσαν για αυτό το θέμα. Είναι ένας τρόπος για να ενημερωθούμε για τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες και ίσως από την ε, μη ορθή εφαρμογή των κανόνων στα κράτη-μέλη. Να τονίσω ότι οι εθνικές αρχές ε, έχουν κάθε δυνατότητα να διοργανώσουν την παροχή δημοσίων υπηρεσιών με όποιον τρόπο θέλουν. Δεν είναι υποχρεωμένες οι δημόσιες αρχές να κάνουν πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών, αλλά αν αποφασίζουν να κάνουν πρόσκληση, τότε δεσμεύονται από την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες. Αλλά ακόμη και αν ένα κράτος μέλος ε, επιλέξει τη διαδικασία υποβολής προσφορών, οι κανόνες που προβλέπει η οδηγία του 2014 αφήνουν πολύ περιθώριο στις εθνικές αρχές, τις δημόσιες αρχές, στα κράτη-μέλη, όχι μόνο να λάβουν υπόψη την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, αλλά επίσης να λάβουν και υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων, των χρηστών αυτών των υπηρεσιών. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ε, προς τα άτομα με αναπηρία. Εδώ υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο και χωριστό ειδικό καθεστώς που παρέχει πολύ νομική ευελιξία και απαιτεί από τις εθνικές αρχές να λάβουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν και την ενδεχόμενη επίπτωση που θα έχει επί των ε, δικαιούχων. Οι οδηγίες αυτές έχουν ε, μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία στις αρχές του τρέχοντος έτους Άρα υπάρχουν όλες τις δυνατότητες που προβλέπουν οι οδηγίες. Αλλά ορισμένες φορές διαπιστώνουμε ως Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι κυρίως ε, η τοπική αυτοδιοίκηση συχνά δεν έχει ας πούμε το αναγκαίο θάρρος για να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που παρέχει το νομικό καθεστώς. Οπότε θεωρούμε ότι ο ρόλος μας τώρα, αλλά και στο μέλλον, θα πρέπει να είναι να στηρίξουμε τις εθνικές αρχές στην οργάνωση των ε, διαδικασιών υποβολής προσφορών να είναι πιο ευαίσθητες, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων των υπηρεσιών που προτίθενται να παράσχουν. Χάρη και στη δική σας παρέμβαση, πρόσφατα επικοινωνήσαμε με τις Εθνικές Αρχές της Φινλανδίας για να διευκρινίσουμε μερικά από τα νομικά θέματα που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών προς με αναπηρία. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στήριξη χρειάζεται περαιτέρω διαβούλευση. Επίσης, Αυτή η νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στα πλαίσια των προτεραιοτήτων μας για τις δημόσιες προμήθειες. Δηλαδή, βεβαίως τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε να ανεβάσουμε την ποιότητα των δημοσίων προμηθειών και να ξεπεράσουμε τη λογική του μειοδότη. Αλλά επίσης θέλουμε να αξιοποιηθούν οι δημόσιες προμήθειες για να επιτύχουμε ορισμένους στόχους πολιτικής, ιδιαίτερα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. για να έχουμε πιο ε, βιώσιμα αποτελέσματα μέσω των δημοσίων προμηθειών. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Μας χαροποιεί γιατί δεν συμβαίνει πάντα το πόσο μας ενθουσιάζουν αυτά που λέει η Επιτροπή. Η δική μας Επιτροπή. Με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμεθα πολύ στενά για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Και τονίζω, είμαστε δύο θεσμοί που συνεργάζονται. Τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να ασκήσουμε πολύ πίεση στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με σωστό τρόπο την νομοθεσία. Θα επανέλθω. Αλλά τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Και τώρα η κυρία ε, στην κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ε, έζησα κάτι παρόμοιο. Ένα άτομο με αναπηρίες όταν βρίσκεται σε ένα κέντρο δημιουργεί ένα σύνδεσμο με το προσωπικό. Είναι ένας πολύ, ισχυρό ένας ισχυρός δεσμός με την νοσοκόμα, με τον φροντιστή του, με όλο το προσωπικό που βρίσκεται στο κέντρο. Ε, όταν οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν αντικείμενο δημοπράτησης, ε, ε, σπάει αυτή η αρμονία και η ασφάλεια την οποία νιώθουν τα συγκεκριμένα άτομα. Οπότε σε τέτοιου είδους δημοπρατήσεις πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, να λαμβάνετε υπόψη και άλλοι παράγοντες, όχι μόνο το κόστος οι υπηρεσίες ε, είτε αφορούν άτομα με αναπηρία είτε αφορούν ηλικιωμένα άτομα, άτομα που εξαρτώνται, εξαρτώμενα άτομα δηλαδή γενικά, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλους κοινωνικούς παράγοντες, όχι μόνο το κόστος. Οπότε την εποχή που συζητούσαμε την οδηγία αυτή ως κυβέρνηση των Βαλεαρίδων προσπαθήσαμε ήδη τότε με τροπολογίες που είχαν προτείνει να ευαισθητοποιήσουμε την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Και, η, οδηγία, και το, η Κομισιόν πράγματι το έκανε, γιατί η οδηγία περιλαμβάνει τέτοιες διατάξεις. Το κράτος μέλος όμως θα πρέπει να τις εφαρμόζει σωστά. Οπότε έχω την εντύπωση ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η οδηγία Οπότε αυτό το οποίο είναι προφανές, το ότι δηλαδή αλλιώς ε, δημοπρατούμε τις, υποχ... Ε, υπηρεσίες καθαρισμού και αλλιώς τις κοινωνικές υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό το οποίο είναι λοιπόν προφανές δεν ε, πραγματοποιείται. Η οδηγία το προβλέπει, δίνει περιθώριο, όμως το περιθώριο αυτό δεν το εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οπότε προτείνω να απευθυνθούμε σε συνεργασία με την Κομισιόν σε αυτό το κράτος μέλος για να μας εξηγήσει από μια μεριά και από την άλλη μεριά να το εξηγήσουμε ότι δεν μπορεί να πράττει αυτό που πράττει και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ποιοτικά και κοινωνικά κριτήρια. Όλα αυτά συμβαδίζουν με αυτά που μας είπε και η Κομισιόν. Οπότε ας επευθυνθούμε στην Φιλανδία να μας εξηγήσει τι κάνει και να επιμείνουμε έτσι ώστε να αλλάξει η Φιλανδία αυτές τις πρακτικές των δημοπρατήσεων. Κάθε πέντε χρόνια λένε ε, αλλάζει ο πάροχος, άλλες φορές ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων, άλλες όχι. Οπότε είναι προφανές ότι δεν μπορεί το κόστος να είναι το μοναδικό κριτήριο. Η οδηγία δίνει περιθώριο να σταθμιστούν και άλλα κριτήρια. Οπότε το θέμα είναι θέμα εφαρμογής. Ευχαριστώ. Thank you, Ross. Κυρία Κούλενεν. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που η έχουμε τόσους Φιλανδούς ε, που είναι διατεθειμένοι να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογένειών τους. Να προασπίσουν τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, που δεν έχουν φωνή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπούνται από ομάδες ε, και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ως Φιλανδή Ευρωβουλευτής μπορώ να σας πω ότι είμαι πρόθυμη να στραφώ εναντίον της ίδιας της χώρας μου, διότι είναι ε, κάκιστος ο τρόπος με τον οποίο η Φιλανδία φέρεται στα άτομα με αναπηρίες. Δεν έχουν δικαίωμα μέσω διοικητικής απόφασης να μετακινούν από ε, ένα ίδρυμα σε ένα άλλο τα άτομα αυτά. είναι φυσιολογικό να έχουμε τόσες αναφορές και τόσα παράπονα. Έχουμε εκατοντάδες άτομα που απευθύνονται σε μας και μας καταγγέλουν τέτοιες περιπτώσεις. Δυστυχώς οι κρατικές προμήθειες και οι δημοπρατήσεις ε, θεωρούν τα άτομα με αναπηρίες ε, ως ένα ακόμα γρανάζι ενός μηχανισμού. Δεν τους αναγνωρίζουν κάποια ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όμως, δεν μπορεί να συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως αποστολή να προσπίζει τα άτομα που είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε υφίστανται και οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. προκαλούμε τεράστια οδύνη στα άτομα αυτά και ενδεχομένως και μίσος πολλές φορές. Αυτά τα άτομα πολλές φορές λαμβάνουν ε, φαρμακευτική αγωγή και μερικές φορές χρειάζεται και να τα δέσουν στα κρεβάτια τους, να τα κινητοποιήσουν. Καταλαβαίνετε τι έχουμε τι κατάσταση έχουμε δημιουργήσει. Εγώ έχω δουλέψει ίδια με άτομα, ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες για έξι μήνες σε ένα ίδρυμα ηλικιωμένων και θυμάμαι το πώς είχα χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αλλάξει όλο αυτό, να αλλάζει κάθε πέντε χρόνια για την ακρίβεια, όλο αυτό το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν οι ανάπηροι. Τα άτομα τα οποία τους φροντίζουν ε, φτάνουν στο σημείο να αναγνωρίζουν και το τι σημαίνει η παραμικρή χειρονομία ή το η παραμικρή κίνηση των ματιών και μέσω αυτών επικοινωνούν. Δεν είναι δυνατόν να τους αλλάζουμε κάθε τόσο. Και είναι ντροπή να δεχόμαστε έμεσα το ξεπούλημα των πιο ευάλωτων ατόμων κάθε πέντε χρόνια. Είναι τα άτομα τα οποία που έχουν τη λιγότερη, τη μικρότερη δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους και τα δικαιώματά τους. Αυτό σίγουρα κάπου δείχνει ότι κάνουμε λάθος. Η οδηγία πλαίσιο δεν το απαιτεί, δεν απαιτεί από τη Φιλανδία να λαμβάνει υπόψη μόνο το κόστος των υπηρεσιών αυτών. Οπότε εμείς ως Κοινοβούλιο αλλά και η Κομισιόν μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι αυτό είναι λάθος. Thank you very much. Ευχαριστώ κυρία Κιούλανεν, λέει η πρόεδρο. Και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή. Δεν σα είχα ξαναδεί στο παρελθόν. Σα χρειαζόμαστε να ξανάρθετε. Η κυρία Στανόκα, ω τελευταία ομιλήτρια. Έχοντα ακούσει την απάντηση της Κομισιόν, και βλέποντας το πώς η οδηγία ε, εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη. Μήπως ε, θα έπρεπε η υπόθεση αυτή να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Η Φιλανδία είναι προφανές ότι εφαρμόζει λανθασμένα την οδηγία. Οι αναφερόμενοι μας περιέγραψαν αυτή την ε, κάκιστη κατάσταση. Αλλά εμείς δεν έχουμε νομική βάση για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε μόνο από την Κομισιό να ε, ενθαρρύνει το κράτος μέλος να διορθώσει την κατάσταση. Αλλά παρόλο που δεν είμαι δικηγόρο και δεν γνωρίζω πολύ καλά την οδηγία, δεν υπάρχει περιθώριο προσφυγή στο δικαστήριο. Ίσως κάποιο ε, πιο αρμόδιος θα μπορούσε να με ενημερώσει. Πρόεδρο, κύριε Στανόκα, το καλό είναι ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Φιλανδίας είναι εδώ και είμαι σίγουρος ότι σημειώνει τα όσα λέμε. Όλοι είχαμε την εικόνα ότι η Φιλανδία είναι στην κορυφή και μας εκπλήσει και μας ευνηδιάζει το πόσο το που βρίσκεται η κατάσταση εκεί. Οπότε η μόνιμη αντιπροσωπεία της Φιλανδίας είμαι σίγουρη πως ε, καταγράφει τα σχόλιά μας. Ο χρόνος μας πιέζει. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, αναφέροντες για δύο λεπτά. Εσείς ε, αποφασίστε ποιος θέλετε να πάρει το λόγο. Δεν χρειάζεται να παρουσιάσετε κάποιο καινούριο δεδομένο. Δύο λεπτά για να κλείσουμε απλώς τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όπως ε, σας είπα ήδη, Όλες οι οργανώσεις για τα άτομα με αναπηρίες έχουν ε, προωθήσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών προκειμένου να αλλάξει η νομοθεσία στη χώρα μας, στη Φιλανδία. Και μάλιστα μας δόθηκε και το πράσινο φως από τους υπεύθυνους ανάληψη αποφάσεων σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή. Αυτό το οποίο όμως ε, θέλουμε να ακούσουμε και στα πλαίσια της συζήτησης που θα γίνει την ερχόμενη άνοιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει με την κοινοτική νομοθεσία. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι είναι η κοινοτική νομοθεσία που δεν θα επιτρέψει στι αρμόδιε εθνικέ αρχέ Φιλανδία να επιφέρουν τι αλλαγέ τι οποίε εμεί θέλουμε να δούμε. Απευθύνομαι σε εσά λοιπόν, στην Επιτροπή Αναφορών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλε οι υπόλοιπε αρμόδιε αρχέ για να μα βοηθήσετε. Σα δώσαμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία όλα καταδεικνύουν ξεκάθαρα για το πώς έχει η κατάσταση. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν στη Φιλανδία. Η κατάσταση είναι μη βιώσιμη, ιδίως όσον αφορά τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες. Και η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή πραγματικά απειλεί την ομαλή ζωή και των ίδιων των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο για να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για όλες αυτές τις τρομακτικές ιστορίες που ζούμε στη Φιλανδία. Ο καθένας πάντως από εμά ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι ευθύνε που έχει σε σχέση με τα παιδιά του και που ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για το μέλλον των παιδιών μας προφανώς, ξαφνικά αισθανόμαστε εντελώς αδύναμοι μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, μπροστά στις αποφάσεις που λαμβάνονται για μας χωρίς εμάς. Να λοιπόν το βασικό μήνυμα το οποίο θα ήθελα να προωθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Όταν μιλάω σε Φιλανδούς, δεν είμαι σίγουρη. Περισσότερο με καταλαβαίνετε όταν μιλάω σου ειδικά, έτσι δεν είναι. Αλλά συνήθω μιλάω αγγλικά εδώ πέρα στην Επιτροπή Αναφορών και μάλλον θα συνεχίσω στα αγγλικά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε αυτό το ταξίδι μέχρι εδώ, μέχρι τι Βρυξέλλε, για να θίξετε το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και εκτιμούμε πραγματικά πάρα πολύ τη συμβολή σα. Είμαι πεπισμένη ότι ε, κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την κατάσταση τη δική σας και των οικογενειών σας, αλλά για το σύνολο της χώρας σας, και για το σύνολο της Ευρώπης θα έλεγα. Γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη είναι τόσο σημαντική τελικά. Πραγματικά αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε. Το ζήτημα αυτό είναι ευρωπαϊκής διάστασης. Και οι ομάδες υποστήριξης των απείρων στην Σουηδία, και χαίρομαι πάρα πολύ που τις αναφέρω, λένε ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνετε καμία απόφαση για μας χωρίς εμάς. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρη συμμετοχή τους και των οικογενειών των ανθρώπων με αναπηρία, ή διαφορετικά θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις στο όνομά τους. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκεστε εδώ πέρα σήμερα. Εμείς προφανώς θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή θα αποστείλουμε μια επιστολή, πολύ ισχυρή επιστολή προς τις φιλανδικές αρχές. Θα τις ενημερώσουμε για τη συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα. Θα τις ενημερώσουμε όχι μόνο για την οδηγία του 2014 στην οποία αναφέρεστε, στην αναφορά σας, αλλά θα αναφέρουμε επίσης και την επιπλέον οδηγία που έχουμε, την μεταγενέστερη οδηγία που έχουμε για τις δημόσιες προμήθειες, ο Μάρκ Ταραμπέλα το 2014 επέβαλε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια έκθεση για τη νέα αυτή οδηγία, η οποία αναφέρεται όχι μόνο στο κριτήριο του πιο φτηνού θα έλεγα υποψηφίου, αλλά πέρα από τα οικονομικά κριτήρια αναφέρονται εκεί πέρα και κάποια άλλα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως κριτήρια ποιότητας ή κοινωνικά κριτήρια. Και επίσης θα πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες και κυρίως το άρθρο 19, ένα πολύ σημαντικό άρθρο που αναφέρεται στα ισότιμα δικαιώματα όλων των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ζουν στο πλαίσιο της κοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αν δεν είναι δυνατό αυτό, τουλάχιστον σε ένα φιλικό περιβάλλον. Και να υπάρχει μία συνέχεια στις συνθήκες αυτές διαβίωσης, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί προς το συμφέρον τους. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ουσιαστικά θα πει συμμόρφωση με το δίκαιο. Ξέρετε τώρα ότι στη Φιλανδία η σχετική εθνική νομοθεσία, η οποία επιβλήθηκε όταν στείλατε και εσείς την αφορά του 2015, ανακλήθηκε και αντικαταστάθηκε από μια άλλη νομοθεσία την 1η Ιανουαρίου του 2017. Έχουμε λοιπόν εκεί πέρα μια νέα νομοθεσία η οποία δίνει πολύ σημαντική έμφαση στα κριτήρια εκείνα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα καθώς επίσης και με το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναφέρεται επίσης και στη διαδικασία διαβούλευσης με τους δικαιούχους των υπηρεσιών αυτών, με άλλα λόγια με εσά και με τους συγγενείς σας. Και αυτό θα το τονίσουμε ότι αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται. Και επίσης θα ζητήσω και μία γραπτή απάντηση από τις Φιλανδικές Αρχές προς την Επιτροπή μας. Δεν θα αποστείλουμε λοιπόν απλώς εμείς μια επιστολή και θα του ζητήσουμε να τη διαβάσουν και ενδεχομένω να την οριοθετήσουν. Θα του ζητήσουμε συγκεκριμένα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας. Επίσης, θα ενημερώσουμε την διακομματική ομάδα για την αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα αυτό, καθώ επίση και το EDF, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίε, με το οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Θα του ενημερώσουμε λοιπόν για την αναφορά αυτή και θα απευθυνθούμε και στα υπόλοιπα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λέγοντά του ότι θέλουμε να θίξουμε ήδη σε μια συνεδρίαση που θα έχουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι 6 Δεκεμβρίου τα ζητήματα αυτά τα οποία θίγουμε εδώ πέρα σήμερα. Επομένω, θα αναφερθούμε και τότε στη δική σα την αναφορά. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Βλέπω ότι συμφωνούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κανεί δεν θέλει να προσθέσει κάτι, έτσι δεν είναι. Ή δεν θέλετε να προβάλλετε κάποια αντίρρηση στα όσα είπα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ και χαιρετισμού και στη Φιλανδία που είναι μια πολύ σημαντική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την οποία περιμένουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή επιστροφή στη Φιλανδία. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε τώρα στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης, λέει Πρόεδρος. Μάλλον το σημείο 8 έχει αναβληθεί. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 9 της ημερήσία διάταξης. Αναφορά 696 για την ανάγκη νέα ταξινόμηση τη τοπική αστυνομία από το Ιταλικό κράτο. Και έχουμε επίση και την αφορά 93 για την εξίσωση του νομικού καθεστώτο των τοπικών και δημοτικών αστυνομικών δυνάμεων με εκείνο άλλων εθνικών και ευρωπαϊκών αστυνομικών δυνάμεων. Βλέπω κάποιον που φοράει αστυνομική στολή, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι θα πάρετε το λόγο. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στους δύο αναφέροντες. Πέντε λεπτά ο καθένας, ο κύριος Μαρούκινο πρώτος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ευρώπη που μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τις αναφορές μας αυτές και να εισακουστεί η φωνή των 60.000 εργαζομένων στην τοπική αστυνομία της Ιταλίας. Άνθρωποι που είναι παρόντες σε όλους τους δήμους Ιταλίας, ακόμα και σε μικρούς δήμους, όπως στο Ματρίτσε, που είχαμε ένα πολύ σημαντικό σεισμό και όπου οι υπηρεσίες διάσωσης που πρόσφερε η τοπική αστυνομία ήταν πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και που ουσιαστικά είναι άνθρωποι οι οποίοι παρεμβαίνουν σε όλους τους περιοχές εκείνους που έχουμε σημαντικές καταστροφές. Ακόμα λοιπόν και στους μικρότερους δήμους και στα μικρότερα χωριά έχουμε εκπροσώπους της τοπικής αστυνομίας. 60.000 λοιπόν αυτά άτομα που εργάζονται στην Ιταλική τοπική αστυνομία καλύπτουν όλη την επικράτεια της Ιταλίας και τους 8.000 δήμους της χώρας. Και πραγματικά είναι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές είναι παρόντες στις μικρές αυτές τοπικές κοινότητες, εκπροσωπώντας τελικά το κράτος και εκπροσωπώντας την αστυνομία. Τούτο λεχθέντων βλέπω ότι ήδη βλέπετε στις διαφάνειές σας κάποια ονόματα. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί θα αναρωτιέστε. Μα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσία στα πλαίσια της τοπικής αστυνομίας πάντα. Πάνω από 60 θύματα της τοπικής αστυνομίας έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας σε πάρα πολλέ πόλει μεγάλη Ιταλία, επίση πάρα πολλέ πρωτεύουσε Δήμων και γενικότερα στην επικράτεια τη χώρα μου. 60 θύματα. Ο αριθμό είναι πολύ μεγάλο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε από την Ιταλική κυβέρνηση για ποιο λόγο θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να χάουν τη ζωή του εν ώρα εργασία. Και διαρωτόμαστε και κάτι ακόμα. Για ποιο λόγο χάσαν τη ζωή του οι άνθρωποι αυτοί. Ε, πέθαναν, έχασαν τη ζωή τους, γιατί οι ε, συνάδελφοι αυτοί προσπαθούσαν να επιτελέσουν το έργο τους υπερασπιζόμενοι τα θεσμικά όργανα της χώρας, επιβάλλοντας την τάξη, επιβάλλοντας τον νόμο. Και γι' αυτό το λόγο σφαγιάστηκαν πάρα πολλές φορές στους δρόμους της χώρας μου, δέχθηκαν πυροβολισμού σε πάρα πολλές πόλεις της Νοτιού Ιταλίας αλλά και της Βορείου Ιταλίας και κυρίως ε, οι συνάδελφοι αυτοί που χάσαν τη ζωή τους, έχασαν τη ζωή τους γιατί δεν είχαν την απαραίτητη προετοιμασία, προστασία, τον απαραίτητο εξοπλισμό προστασίας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φέραν καν τα κατάλληλα όπλα. Ξέρετε ότι έχουμε μία τοπική αστυνομία 60.000 εργαζομένων που ουσιαστικά καλείται τώρα να καταπολεμήσει ακόμα και την τρομοκρατία. σε χώρους οι οποίοι θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Επί του παρόντος, η τοπική αστυνομία, ή μάλλον ζητάται από την τοπική αστυνομία, να επιτελέσει καθήκοντα διατήρησης ασφάλειας σε μεγάλα αστικά κέντρα. Για παράδειγμα, στο Κολοσσέο. Ξέρετε ότι κανονικά εκεί πέρα έχουμε παρουσία της στρατιωτικής αστυνομίας ή και του στρατού. Ο στρατός που φέρει τα κατάλληλα μυδραβιοβόλα όπλα. Και δίπλα τους τι έχουμε. Έχουμε αστυνόμους της τοπικής αστυνομίας μέσω του Δήμου της Ρώμης, οι οποίοι όμως δεν έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν φέρουν όπλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εκθέτει πάρα πολύ τους συναδέλφους των οποίο η ασφάλεια δεν προστατεύεται. Για ποιο λόγο λοιπόν χάσαν τη ζωή τους, για ποιο... επειδή δεν είχαν την κατάλληλη προστασία, δεν φορούσαν αλεξίσφαιρο γυλαίκο, δεν είχαν τα απαραίτητα όπλα, δεν είχαν καμία απολύτως προστασία. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η πατρίδα μας μαζί με την Ιταλία, να αποδώσει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για τα θύματα αυτά. Και διαρωτόμαστε επίσης για ποιο λόγο για ποιο λόγο άραγε η τοπική αστυνομία της Ιταλίας σε αντίθεση με άλλες τοπικές αστυνομίες που έχουμε σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διαφορετική μεταχείριση. Και διαφορετική μεταχείριση ακόμα και από την κεντρική εθνική αστυνομία. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε μία σύμβαση η οποία ουσιαστικά εξισώνεται με τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δήμων και των κοινοτήτων. Στην πράξη είμαστε διοικητικοί πάλι των Δήμων και των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τη σύμβασή μα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε μία συγκεκριμένη εβδομάδα εργασία. Κάθε μέρα θα έπρεπε να εργαζόμαστε από τι 7 το πρωί στι 2 το μεσημέρι και να επιστρέφουμε στα σπίτια μα, στα Σαββατοκύριακα και να ζούμε μια ομαλή, ευχάριστη ζωή. Δεν συμβαίνει όμω κάτι τέτοιο με του εργαζόμενου τοπική αστυνομία. Εργαζόμαστε εντελώ διαφορετικά ωράρια Εργαζόμαστε επίση και κατά τη διάρκεια των νεορτών, ακόμα και τα Χριστούγεννα, ακόμα και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως ακριβώς δηλαδή και οι αστυνόμοι της Εθνικής κεντρική Αστυνομίας, μόνο που εμείς δεν έχουμε συγκεκριμένη σύμβαση που αναγνωρίζει τα καθήκοντά μας αυτά. Μας επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή καθήκοντα τα οποία θα έπρεπε τελικά να αντικατοπτρίζονται κάπω και σύμβασή μα. Εμεί ε, είμαστε υπερήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε. Θέλουμε πραγματικά να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε. Θέλουμε να κάνουμε την επιπλέον αυτή δουλειά που μα ζητείτε αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλουμε να έχουμε και το απαραίτητο προστατευτικό πλαίσιο. Θα πρέπει να έχουμε την κατάλληλη κατάρτιση, την κατάλληλη προετοιμασία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε όλε αυτέ τι νέε απειλέ που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Και όχι μόνο αυτό για να εργαζόμαστε εμείς καλύτερα, αλλά για να μπορούμε πραγματικά να προσπιζόμαστε καλύτερα τους κατοίκους των ε, πόλεων, των Δήμων και των Κοινοτήτων της Ιταλίας. Αυτή τη δουλειά επιτελούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη δουλειά αυτή κάναμε ανέκαθεν. Αλλά μοιάζει η δουλειά αυτή να είναι σαν μια δήλωτη δουλειά αυτή τη στιγμή. Πρόεδρος, ε, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνο αγόρευση που είχατε και πραγματικά για να δώσουμε και τη δυνατότητα στον αδελφό να πάρει το λόγο, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω, Πρόεδρε. Ολοκληρώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή σας και ζητώ για μία ακόμη φορά μέσω όλων αυτών των στοιχείων που σας δώσαμε να υπερασπιστείτε την υπόθεσή μας, την αναφορά μας. Θα μπορούσα να μιλήσω για πάρα πολλή ώρα, αλλά ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ωραία. Στον αδελφό σου τώρα έχει το λόγο. Μικρόφωνο σας παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Με την αναφορά μας 93 για την τοπική και δημοτική αστυνομία. Οι αρχές αυτές είναι πολύ κοντά στους πολίτες και είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Ορισμένες δραστηριότητες, ε, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ πέρα, η τοπική αστυνομία ψάχνει με σκύλους για ναρκωτικά και είναι στις ε, παραλίες για την ασφάλεια των πολιτών, είναι, επίσης έχουν καθήκοντα τροχέας και ε, ελέγχουν επίσης τις δραστηριότητες μετανάστευσης και διάσωσης. Είναι επίσης πολιτική προστασία και περιβαλλοντική ασφάλεια. Τι μπορούμε να κάνουμε η τοπική αστυνομία στους Δήμους εργάζεται για να αποφευθεί η ριζοσπαστικοποίηση, η τρομοκρατία και ο εξτρομισμός για ένα μέλλον ειρήνης και ενότητας. Βλέπετε εδώ τις εικόνες. Εδώ αριστερά είναι η ριζοσπαστικοποίηση και η τρομοκρατία και ο εξτρομισμός. Πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά. Η τοπική αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την ανθρώπινη ευφία τη, μάλλον τις πληροφορίες που μας δίνουν οι ανθρώπινες ε, πηγές σε αντιπαράθεση με τις ε, τεχνικές προφορίες ε, μέσω τηλεπικοινωνιών που είναι ακριβή όπως τα ξέρετε, θα πρέπει να θυμάστε ότι οι πληροφοριοδότες, οι ανθρώπινες πηγές ε, πληροφοριών είναι πολύ πιο φτηνές σε αντιπαράθεση με μετρήσεις και παρέμβαση στις τηλεπικοινωνίες ελπίζω να υπάρξει μια νέα επιτροπή για την τρομοκρατία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, ξέρω ότι υπάρχει αυτή η νέα επιτροπή και θα ήθελα να σταλεί εκεί για να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για την τρομοκρατία, την ριζοσπαστικοποίηση, τι ευρωπαϊκέ ε, τοπικέ αστυνομίε και την χρήση ανθρωπίνων πηγών. Εδώ βλέπετε ε, συναδέλφους οι οποίοι φέρουν όπλα, αλλά όπως είπε και ο συναδελφός μου στην Ιταλία, δεν έχουν όλοι οι τοπικοί αστυνομικοί ε, όπλα. Ορισμένες φορές έχουμε βέβαια και τη φέκια. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτή η αναφορά έχει στόχο να υπηρετήσουμε και να προστατεύσουμε καλύτερα τη χώρα μου και την Ευρώπη όπως κάνει η τοπική αστυνομία κάθε μέρα. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να πω. Είναι και αυτό που έγραψα και στην ε, εργασία μου. Ε, για να αποφυτίσω ότι για την ειρήνη χρειάζεται και συγχώρηση. Ε, χρειαζόμαστε και την, ε, τις πηγές πληροφοριών, τη δικαιοσύνη αλλά και την συγχώρηση. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει. Ο κύριος Γοντού και ο κύριος Μαρκέτη. Ευχαριστώ. Θα ασχοληθώ με, το, με την αναφορά 0696 όπως λέει και ο αναφέρον και έχουμε κάθε κατανόηση προς τα θέματα που αφορούν την τοπική αστυνομία. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που παίζει η τοπική αστυνομία για τα θέματα ασφάλειας και για την εγγύηση των κοινωνι... της ειρήνης των κοινωνιών μας και για τους ε, πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Όπως λέει η απάντηση της Κομισιόν, με βάση το νομικό πλαίσιο, όλα αυτά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, συγκεκριμένα της Ιταλίας. Μόνο η Ιταλία μπορεί να αποφασίσει ε, τι καθεστώς θα έχει η τοπική αστυνομία και τι εξοπλισμός, ε, κατάρτιση, καθήκοντα και υποχρεώσεις θα τους δοθούν. Έχουμε λοιπόν κάθε κατανόηση, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία δυνατότητα να πάρει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να μιλήσει και ο κύριος Μαρκέτη. Θα πρέπει να επαναλάβω και για τα θέματα των, της, ε, του επιδόματος ασθενείας και των κοινωνικών επιδομάτων. Όλα αυτά είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε τις ανησυχίες τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομοι. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι. Ο κύριος Βαλέντσα. Ευχαριστώ. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Οι αστυνομικοί αυτοί αντιμετωπίζουν πολλούς κινδύνους θα έπρεπε να τους παρέχεται οποιαδήποτε δυνατή προστασία και κοινωνικές παροχές και από πλευράς εξοπλισμού. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από αυτά που λέει η Κομισιόν. Να στείλουμε μια επιστολή στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επιτροπή συνταγματικών θεμάτων, για παράδειγμα. Και να τους παρακαλέσουμε να επανεξετάσουν ε, το καθεστώς Τη τοπική αστυνομία και μπορούμε να στείλουμε επιστολή και στον Υπουργό Εσωτερικών να περιγράψουμε την κατάσταση και να ζητήσουμε τη γνώμη του, να το ζητήσουμε να επανεξετάσει το καθεστώς της τοπικής αστυνομίας. Και επίσης να ρωτήσουμε και τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχουμε τώρα και την Επιτροπή για την Τρομοκρατία. Ας ε, απευθυνθούμε και σε αυτές τις επιτροπές. Υπάρχουν αυτές οι τρεις δυνατότητες το θέμα αυτό, η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να ε, εξετάσουμε την εξέλιξη της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντανόκα. Δεν θα πω πολλά. Είχα τις ίδιες απόψεις με τον κύριο Βαλέντσα. Να στείλουμε μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές και στους συναδέλφους μας Ίσως θα μπορούσε να εμπλακεί και η Επιτροπή Απασχόλησης. Γιατί υπάρχουν τα θέματα της κοινωνικής προστασίας, τα κοινωνικά θέματα δηλαδή, των επιδομάτων. Στηρίζω πλήρως ε, την αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να επιχειρήσουμε να πείσουμε και τις Ιταλικές αρχές, ακόμη και τις νομοθετικές αρχές να κάνουν κάτι για την τοπική αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εύη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο αναφέροντες οι οποίοι συμμετείχαν σε σημερινή συνεδρίαση που έθιξαν το ζήτημα αυτό το οποίο πραγματικά εισάγει πολύ σημαντικές διακρίσεις, διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα στη δική μου τη χώρα ανάμεσα στην τοπική αστυνομία και τις υπόλοιπες μορφές της κρατικής αστυνομίας. Και καταλαβαίνετε ότι όπως ακούσαμε αυτό εκθέτει ιδιαίτερα τους εργαζομένους της τοπικής αστυνομίας οι οποίοι διατρέχουν πλέον πάρα πολλούς κινδύνους προασπιζόμενοι την ασφάλεια των πολιτών της χώρας. Σαφώς πρόκειται λοιπόν για διακριτική μεταχείριση και αυτό θα πρέπει να τονιστεί. Το κίνημα των πέντε αστέρων και στα πλαίσια της Ιταλίας προσπάθησε να προωθήσει το ζήτημα αυτό, να γύρει το ζήτημα αυτό, αλλά δεν μας δόθηκε καμία απάντηση. Ελπίζω λοιπόν ότι τουλάχιστον δική μα η Επιτροπή, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα μπορέσουμε αν μη τι άλλο να στείλουμε μια επιστολή προς τι Ιταλικέ αρχές. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας το είπε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά της το ζήτημα αυτό. Πάντως θεωρώ το ζήτημα είναι σαφώ πολιτική φύση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν μπορούμε να το επιλύσουμε από μόνοι μα και είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με όλε τι πτυχές του προβλήματος. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε για τι παροχέ κοινωνική ασφάλισης, τι παροχέ οικονομική περίθαλψης, που πρέπει προφανώ να παρέχονται στου ανθρώπου αυτού οι οποίοι διακινδυνεύουν πλέον τη ζωή του όλο και περισσότερο, ιδίω στα πλαίσια τη μεγάλη κρίση που ζούμε και κυρίω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Κύριο έχει το λόγο. Σύριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μα προφανώς και εγώ συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους μη Ιταλούς συναδέλφους οι οποίοι ε, μας υποστηρίζουν ε, στις απαιτήσει μας. Μια κατάσταση την οποία γνωρίζω πολύ καλά γιατί εγώ ήμουν επίτροπος και ελεγκτής για ζητήματα τοπικής και δημοτικής αστυνομίας ε, στα πλαίσια του Δημοτικού, Δημοτικού Συμβουλίου της δικής μου της πόλης. Είχα ασχοληθεί λοιπόν με το ζήτημα αυτό και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την σημαντική δουλειά που κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε εμεί δεν έχουμε άμεση αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό. Είπε όμω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το αίτημα των εκπροσώπων της τοπικής αστυνομίας. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και επ' αυτού νομίζω ότι μπορούμε όντω να συντάξουμε μία επιστολή ή να προχωρήσουμε σε μία δήλωση, σε μία ανακοίνωση που θα μπορούσε να πάει και στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και στην Ιταλική Γερουσία. Ξέρετε ότι άλλωστε είναι το Ιταλικό Κοινοβούλιο που ασχολείται με το καθεστώς αυτό της τοπικής αστυνομίας. Πρώτον, το ζήτημα αυτό δεν θα πρέπει πραγματικά να ξεχωρίζει την Ιταλία από τις υπόλοιπες χώρες. Αν πραγματικά θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να λειτουργεί με τρόπο ευθυγραμμισμένο, θα πρέπει ευθυγράμμιση να υπάρχει και στο ζήτημα αυτό. Δεν είναι λογικό ούτε αποδεκτό να, να προστατεύεται λιγότερο ένας αστυνόμος της τοπικής αστυνομίας της Ιταλίας σε σχέση με έναν αστυνόμο από το Βέλγιο, τη Γαλλία ή κάποια άλλη χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι στην επιστολή μας, κυρία Πρόεδρε, θα μπορούμε και αυτό να το λέμε, να πούμε ότι και το Φεβρουάριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε μια πολύ σημαντική δήλωση όσον αφορά την τρομοκρατία. Κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνάμεις οι αστυνομικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Και βέβαια, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να αφήνουμε εκτεθειμένους τους άνδρες και τις γυναίκες της Ιταλικής τοπικής αστυνομίας, οι οποίοι όπως ακούσαμε δεν έχουν ούτε χέγγια ούτε συγκεκριμένη προστασία. Η δράση τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πολύτιμη η Ιταλική τοπική και δημοτική αστυνομία προφανώς θα πρέπει να εξισωθεί σε σχέση με τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αστυνομικές δυνάμεις της χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Απευθύνουμε εκ νέου στους αναφέροντες. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να σχολιάσετε πολύ σύντομα, πολύ σύντομα τα όσα ακούσατε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους ευρωβουλευτές οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί μαζί μας. Όντως, πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι θα πρέπει να αποτανθούμε στις εθνικές αρχές και στις κυβερνήσεις. εδώ μιλάμε για δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε απλώς για ζήτημα δημόσια τάξης ή ασφάλειας. Ζητήματα που προφανώς τα διευθετεί το κράτος, το εθνικό κράτος. Εδώ μιλάμε για ζωές, για δικαιώματα. Μιλάμε για ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους σαν ώρα εργασίας. Ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Ο καθένας βέβαια επιτελεί την εργασία του. Εμείς το μόνο το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρουμε να επιτελούμε καλύτερα το έργο μας. Τα παιδιά μας φοιτούν σε σχολεία πολυπολιτισμικά. Όντως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πως έχουν τα πράγματα. Ακούνε πάρα πολύ συχνά αυτό το οποίο συμβαίνει τελικά στην Ιταλία. Ενημερώνονται για τόσα συμβαίνουν. Ενημερώνονται από εμά, ενημερώνονται από όλη την τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε λοιπόν πράγματι να συμβάλλουμε στην επιβολή του νόμου αλλά και στην προστασία από τρομοκρατία αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο, με την πλαισίωση αυτή δηλαδή, ώστε να μην χάνουν τη ζωή τους οι συνάδελφοί μου. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν σας ε, ζητούμε να επέμβετε για τους 60.000 αυτούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν προστατεύονται οι άνθρωποι αυτοί, αυτό αποτελεί από μόνο του έγκλημα πραγματικά. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά που κάνετε το ταξίδι μέχρι τις Βρυξέλλες και που ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Επιτροπή μας για το πώς έχει κατάσταση και το σύνολο της Ευρώπης βέβαια για το πώς έχει κατάσταση στη χώρα σας. Να κάνω κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Στην όμως ήταν και ο πατέρας μου. Επομένω, καταλαβαίνετε το ζήτημα αυτό με αφορά όλου ιδιαίτερω. Από προσωπική πλευρά πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και από προσωπική πλευρά που θίξετε το ζήτημα αυτό και που ήρθατε να μα μιλήσετε για το ζήτημα αυτό εδώ στι Βρυξέλλε. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Θα στείλουμε μια πολύ άμεση, αν θέλετε, ειλικρινέστατη επιστολή προ τι Ιταλικέ αρχέ, όπου θα αναγνωρίζουμε εκεί ότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές επιτελούν ένα καταπληκτικό έργο και ότι αποτελούν πάρα πολύ σημαντικούς εταίρους της κοινωνίας σε πάρα πολλούς τομείς. Και θα εξηγήσουμε επίσης στις Ιταλικές αρχές ότι ε, η απόκληση που υπάρχει ανάμεσα στην τοπική αστυνομία και στους ε, αστυνόμους κεντρικής αστυνομίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αφενός δημόσιες συμβάσεις και από την άλλη συμβάσεις ιδιωτικής φύσης. Όπω έχει πει όμω και στο παρελθόν, ήδη από τον Οκτώβριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ιταλία είναι η μόνη αρμόδια για τι κοινωνικέ τη πολιτικέ, για το σχεδιασμό και την διαχείριση των πολιτικών αυτών. Αναγνωρίζουμε προφανώ το γεγονό αυτό, αλλά λέμε παράλληλα ότι η Ιταλία θα μπορούσε να πάει και πολύ καλύτερα, ότι θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό αξίζει να τονίσουμε, πιστεύω, προ Ιταλικέ αρχέ. Και όπω είπε ο συνάδελφο Βαλέσα, θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να θεωρήσουν το εφιστάμενο πλαίσιο, να τροποποιήσουν το πλαίσιο αυτό και να παράσχουν πιο ισότιμες και δίκαιες συνθήκες για τους εργαζόμενους της τοπικής αστυνομίας, οι οποίοι εργάζονται και αυτοί προς το όφελος της κοινωνίας. Και στο τέλος της επιστολής αυτής θα λέμε ότι η δική μας η Επιτροπή, η Επιτροπή των Αφορών, υποστηρίζει τα αιτήματα των αναφερόντων. Και θα πούμε για μία ακόμη φορά ότι ως φίλοι βασικά της Ευρώπης θεωρούμε ότι η Ιταλία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος μέλος και θα πρέπει ουσιαστικά να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα. Θα πρέπει να βελτιώσει επιδόσεις της. Ας το θέσουμε κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν θα πράξουμε και θα στείλουμε επίση και μια ενημερωτική επιστολή όπως το ζήτησαν και οι συνάδελφοι προ την Επιτροπή Απασχόλησης και προς την νέα ειδική επιτροπή, προσωρινή επιτροπή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφέρομαι στην Επιτροπή ΤΕΡ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να αποστείλουμε μια επιστολή αν το επιθυμείτε. Πάντω νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρα πολλά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή Τρομοκρατίας, άρα θα μπορούσε να ασχοληθεί και με το ζήτημα αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να ασχοληθούμε έτσι και περαιτέρω με το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να σκηνηθούμε έτσι. Για άλλη μια φορά σα ευχαριστώ πολύ που ταξιδέψετε μέχρι τι Βρυξέλλες, που είστε εδώ πέρα σήμερα. Σα εύχομαι μια ευχάριστη επιστροφή, καλή επιστροφή στην όμορφη Ιταλία. Αγαπητοί συνάδελφοι, α περάσουμε τώρα στο σημείο 10 τη ημερήσια διάταξη. για το θέμα των υποτιθέμενων παραβιάσεων της Ιαπωνίας στο Διεθνές ε, ε, Μορατόριουμ για την ε, Φάλαινα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία Ελεύθερων, Ελεύθερων Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φέντερ, τον αναφέροντα, για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που δίνετε στην οργάνωσή μας στην WDC το λόγο. Το Μάρτιο του 2014 το πρόγραμμα ε, αλίας ε, της Ιαπωνίας για τις φάλαινες στον Ανταρκτικό ωκεανό κηρύχθηκε παράνομο γιατί δεν γίνεται για επιστημονικούς λόγους από το Διεθνές Δικαστήριο. Ε, Παρ' όλα αυτά τον Οκτώβριο 2015 η Ιαπωνία δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από την δικαιοδοσία του Διεθνούς ε, Δικαστήριου ε, ζητώ συγγνώμη του διακόπτη πρόεδρος. Πρέπει να ζητήσω από τους Ιταλούς φιλοξενούμενους να μην κάνουν θόρυβο. Παρακαλώ πολύ συζητήστε εκτός της αιθούσης. για να συγκεντρωθούμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ πολύ μπορείτε να βγείτε εκτός εθούς ή να συνεχίσετε. Παρακαλώ συνεχίστε. Παρ' όλα αυτά, τον Οκτώβριο του 2015 η Ιαπωνία δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την ε, επιστημονική αλίευση της ε, φάλαινας. Το Νοέμβριο 2015 η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει ε, την αλίευση φάλαινας στον Ανταρκτικό μέσω του προγράμματος New Rep Alpha παρόλο στις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και την συνολική αντίδραση. Στόχος του σχεδίου ήταν να θανατωθούν 4.000 φάλαινες στα επόμενα 12 χρόνια, 333 ανά έτος. Ε, η Διεθνής Επιτροπή ε, για τη Φάλαινα ε, υιοθέτησε δύο ψηφίσματα, το 2014 και το 2016, αναφέροντας ότι δεν μπορούν να εκδοθούν άλλες άδειες αλίευσης για επιστημονικούς λόγους μέχρι ότου η Επιστημονική Επιτροπή του IWC είχε επιβεβαιώσει ότι είναι για επιστημονικούς λόγους. Όμως αυτή η Επιτροπή ε, ότι το πρόγραμμα New Rep A της Ιαπωνίας δεν πληρεί τα κριτήρια για να θεωρηθεί ότι είναι επιστημονικό πρόγραμμα. Από το 2015 η Ιαπωνία έχει θανατώσει 666 φάλινες ε, ε, στο πλαίσιο του πρόγραμματος New Rep Α. Τον Νοέμβρη του 2016 η Ιαπωνία εισήγαγε το πρόγραμμα New Rep NP για ένα νέο πρόγραμμα στο Βόρειο Ειρηνικό με στόχο να ξεκινήσει αλίευση από το 2017 για 130 τέσσερις Σάι Μίνκι και Σάι ε, Wales και 170 Μίνκι φάλαινες κατέτος για 12 έτη. Και πάλι η Επιτροπή Φαλαινοθυρίας δεν στήριξε την Ιαπωνία ε, και δεν επιβεβαίωσε την για επιστημονικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, στις 3 Νοεμβρίου 2017 η Ιαπωνία ξεκίνησε την περίοδο αλίευσης στο Βόρειο Ειρηνικό με 134 Σάι και 128 μην κυφάλαινες να θανατώνονται. Το 2017 το Κοινοβούλιο του, της Ιαπωνίας ε, συμφώνησε ένα νέο νόμο ε, για να ξεκινήσει η εμπορική αλήψη φάλαινας. Επιπλέον, η οι πράξεις αυτές της Ιαπωνίας παραβαίνουν την διαδικασία της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθυρίας και τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά επίσης και τη σύμβαση του Διεθνούς Εμπορίου για τα ε, είδη που απειλούνται, τις ΣΥΤΕΣ. Ε, η Ιαπωνία ε, το, το παράρτημα της ΣΑΙΤΣ και η Ιαπωνία δεν έχει υποβάλει επιφύλαξη για το Βόρειο Ειρηνικό. Από το 2002 η, η Ιαπωνία έχει θανατώσει 1.400 φάλαινες σε διεθνή ύδατα. Επιπλέον, η παραβίαση της ΣΥΤΕΣ ε, συζητείται ε, αυτή τη βδομάδα στην Γενέβη από την, Επιτροπή, από τη μόνη Επιτροπή της ΣΥΤΕΣ. Στην εισαγωγή στην Οικονομική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-Ιαπωνία σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε ό,τι αφορά τις διεθνείς υποχρεώσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία δεσμεύονται να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις ε, υποχρεώσεις τους σε ένα πολυμερές ε, περιβάλλον συμφωνιών. Ε, η Διεθνή Σύμβαση για την Φαλαινοθυρία είναι μια τέτοια συμφωνία. Επιπλέον, η ΣΥΤΕΣ αναφέρεται ρητά στο έγγραφο, όπως είπαμε και προηγουμένως. Η Ιαπωνία συνεπώς παραβαίνει σαφέστατα την ε, απαγόρευση της ΣΥΤΕΣ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρές πολιτικές εναντίον τι φαλαινοθυρίε, είτε είναι εμπορική είτε είναι επιστημονική. Ε, την τελευταία δεκαετία έχει αναφερθεί, έχουν αναφερθεί επανειλημμένω οι ανησυχίε τη Ιαπωνία ό,τι αφορά τα δίθεν επιστημονικά προγράμματα τη Ιαπωνία. Επιπλέον, το 2012 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο σημείωσε ότι σημαντικέ διαφοροποιήσει παραμένουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιαπωνία σε θέματα σχετικά με την διαχείριση τη αλία και τη φαλαινοθυρία, ιδιαιτέρω την φαλαινοθυρία εκ μέρους της Ιαπωνίας ε, ε, ε υπό την ε, ε υποτιθέμενη επιστημονική της δράση ενώ το 2016 το ψήφισμα του πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει με την Ιαπωνία για μια στρατηγική συμφωνία εταιρική σχέση και μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και κάλεσε την Κομισιόν, την Υπηρεσία Εξωτερικής δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να πιέζουν την Ισπανία για το θέμα τη ε, υποτιθέμενης ε, επιστημονική φαλαινοθυρία, προκειμένου να καταρριφθεί αυτή η πρακτική χρησιμοποιώντα πολυμερή και διμερή κανάλια. Το 2017 σε άλλο ψήφισμα για την φαλαινοθυρία στην Νορβηγία το Κοινοβούλιο Συμβούλιο επίση ανέφερε ότι το αυξανόμενο εμπόριο προϊόντων φαλαινοθυρία μεταξύ Νορβηγίας και Ιαπωνία υποσκάπτει την, τον κανονισμό τη ΣΥΤΕΣ. Αντιθέτως με αυτό πιστεύει η Κομισιόν, εμεί είμαστε ε, Θεωρούμε, είμαστε πεπισμένοι ότι οι διαπραγματεύσει, ε, οι τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πιεστεί η Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι θα χρησιμοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που διαθέτει προκειμένου να φέρει σε πέρα στις ευθύνε που έχει αναλάβει. Αν όχι, το ευρωπαϊκό κοινό δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ε, παραδεχτεί ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές διατήρησης ε, ε, υπόκεινται σε οικονομικά κριτήρια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Στρέφομαι στους εκπροσώπους της Κομισιόν, ο κ. Ρισίρ και ο κ. Κυρούλου. Thank you very much, uh, Madam Chair. On Εκ μέρους της Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την, το ότι εκφράζει το τα, τις ανησυχίες πολλών Ευρωπαίων πολιτών, ε, θεμητές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως προσιλωμένη στην ε, διατήρηση όλων των ειδών της ΣΥΤΕΣ. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπεται η εμπορική φαλαινοθήρια. Επίσης δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και εξαγωγή τέτοιων ειδών. Σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως έχει υποστηρίξει το Παγκόσμιο Μορατόριο της ε, Εμπορικής Φαλαινοθυρίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθυρίας και έχουμε τεθεί κατά της εμπορίας τέτοιων ειδών στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΣΥΤΕΣ. Ε, Δραστήρια έχουμε εκφράσει την αντίδρασή μας ε, ε, κατά της φαλαινοθυρίας εμπορικής ή επιστημονικής εκμέρωσης της Ιαπωνίας. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσόρισε την απόφαση του διεθνού Δικαστηρίου που ε, διέτασε την πάυση του πρόγραμματος φαλαινοθυρίας Ιαπωνίας και το 2015 διπλωματικά ε, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία και την ε, Αυστραλία καταγγείλαμε την ε, Ιαπωνία το 2016 στο πλαίσιο της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθυρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε την υιοθέτηση ψηφισμάτων που, που διευκρίνιζαν την χορήγηση επιστημονικών αδειών ε, την όλη διαδικασία και τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίως εξέφρασε τις ε, σημαντικές ανησυχίες που έχει σε ό,τι αφορά τη χρήση εκ μέρους Ιαπωνίας των επιστημονικών προγραμμάτων φαλαινοθυρίας. Ε, καθώς επίσης καταγγείλαμε και την φαλαινοθυρία φαλαινών ΣΕΙ από την Ιαπωνία που ε, όλα αυτά αποδεικνύουν όμως ότι ε, η στάση μας αυτή δεν οδήγησε στη χαλάρωση ε, εκ μέρους της Ιαπωνίας, της στάσης της. Η, αντιθέτως, η Ιαπωνία ε, ε, απέσυρε τις περιοχές φαλαινοθυρίας από τις περιοχές στις οποίες δέχεται την δικαιοδοσία του Εθνούς Δικαστηρίου, δηλαδή σκλήρινε τη στάση της. Ε, το να χρησιμοποιήσουμε τι εμπορικέ διαπραγματεύσει για να πιέσουμε την Ιαπωνία σε ό,τι αφορά τη φαλαινοθυρία μπορεί να έχει ευρύτερε αρνητικέ επιπτώσει στι διμερεί σχέσει. Αλλά επιπλέον αμφιβάλλουμε για το κατά πόσον αυτό θα μα βοηθούσε να πετύχουμε το στόχο μα σε ό,τι αφορά δηλαδή την πάυση τη φαλαινοθυρία. Επίση, ενδεχομένω κάτι τέτοιο θα μείωνε τι ευκαιρίε που έχουμε να συζητούμε διμερώ με την Ιαπωνία για άλλου είδου ε, περιβαλλοντικά ζητήματα. Τούτου λεχθέντος. Η μια ε, εμπορική συμφωνία που θα μας διευκόλυνε να ε, διευρύνουμε τη σχέση μας για περιβαλλοντικά θέματα θα ήταν καλή. Ε, στο πλαίσιο της σύμβασης της ΣΥΤΕΣ αυτό μπορεί να γίνει και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Όμως χρειάζεται αμοιβαία αποφασιστικότητα και επιθυμία. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα συνεχίσουν ε, να θίγουν το θέμα αυτό σε, διμερή, σε και πολυμερή φόρα. Και να σας πω τα εξή δύο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ε, συμμετέχει στη μόνιμη επιτροπή της ΣΥΤΕΣ και εκεί πιέζουμε την Ιαπωνία να συμμορφωθεί σε ό,τι αφορά τον Βόρειο Ειρηνικό και την αλίευση εφαλινών ΣΕΙ. Σήμερα το πρωί μάθα ότι ως αποτέλεσμα αυτής της πίεσης η Ιαπωνία αποφάσισε να δεχθεί επίσκεψη της γραμματείας της ε, ε, Μόνιμης Επιτροπής ΣΥΤΕΣ που θα ερευνήσει τις ε, απαντήσεις που έχει δώσει η Ιαπωνία ε, για τη φαλαινοθυρία. Αυτό τους επόμενους μήνες. Προφανώς δεν αρκεί, δεν αρκεί αυτό, αλλά είναι ένα καλό πρώτο Δεύτερον, το Σεπτέμβριο η Επιτροπή υπέβαλε την ε, πρότασή της για την ευρωπαϊκή θέση για τις επόμενες τρεις ε, συνεδριάσεις της, Ευρωπαϊκής, της Επαγκόσμιας Επιτροπής, ε, Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθυρίας. Ε, ε, εκεί επιβεβαιώνουμε ότι η Κομισιόν υποστηρίζει την συνέχιση του μορατόριου ε, και μια διαδικασία, διαφανή διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό για τώρα και για τα επόμενα χρόνια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει προσιλωμένη στην ε, διατήρηση των ειδών της προστατεύονται από τις ΣΥΤΕΣ. Και θα συνεχίσουμε να θίγουμε το θέμα της φαλανοθυρίας εκ μέρους Ιαπωνίας. Ευχαριστώ. Good morning. Um, Καλημέρα. Όπως μόλις είπε ο συνάδελφός μου, η Επιτροπή κάνει διάφορες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το θέμα σε όλα τα δυνατά βήματα. Βεβαίως έχουμε το κεφάλαιο του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης και θα αποτελέσει τμήμα της συμφωνίας μας με την, Ένωση, με την Ιαπωνία. Είναι ένα επιπλέον βήμα για να υπάρξει διάλογος μεταξύ Ένωσης και Ιαπωνίας για περιβαλλοντικά θέματα που έχουν σχέση με τις εμπορικές σχέσεις. και για την φαλαινοθυρία και για την εισαγωγή κρέατος φάλαινας. Όπως σας είπα αυτά και τα δύο απαγορεύονται στην Ένωση. Οπότε για μας δεν δείτε θέμα. Δεν είναι θέμα η φαλαινοθυρία. Δεν είναι θέμα εμπορίου. Δεν είναι θέμα το οποίο υπάγεται στην εμπορική μας πολιτική. Αλλά έχουμε, όπως είπα, κάποιες δυνατότητες να θίξουμε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού. Αλλά σύμφωνα με την ε, εσωτερική μας αξιολόγηση, αν επιμείνουμε ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Τι δυνατότητες έχουμε εντός της εμπορικής πολιτικής. Αυτές έχουμε και με αυτές προσπαθούμε να πορευτούμε στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου που ανέφερα. Και στο κεφάλαιο αυτό αναφερόμεθα και στη συμφωνία ΣΥΤΕΣ. Ευχαριστώ. Κυρία Μινά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον αναφέροντα της οργάνωσης αυτής ε, WDC και τις 276.000 ε, υπογράφοντες. Στηρίζω το αίτημά τους. Οι φάλαινες ε, απειλούνται σοβαρά και έχει υπάρξει ένα μορατόριο στη φαλαινοθυρία από το 1982. Το κρέας της φάλαινας δεν καταναλώνεται τόσο πλέον στην Ιαπωνία. Εκατοντάδες φάλαινες δολοφονούνται κάθε χρόνο χωρίς κανένα λόγο και λαμβάνει επιδότηση ο κλάδος. Και το πρόσχημα της Ιαπωνίας είναι ότι γίνεται για επιστημονικούς λόγους. Το 2016 το Κοινοβούλιο επέμεινε έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών να γίνει οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει για να επιλυθεί το θέμα αυτό μέσω πολιτικού διαλόγου. Και ζητήσαμε να, να υπάρξει η μέγιστη δυνατή βιώσιμη ανάπτυξη και σε τομείς όπου δεν υπάρχει εμπόριο. Η Κομισιόν δεν χρειάζεται και δεν βοηθάει να ασκήσουμε πίεση στην Ιαπωνία. Αλλά ξέρουμε ότι η Ιαπωνία έχει αποσύρει τις αντιλήσεις της για την ε, ε, απαγόρευση της εμπορικής ε, φαλινοθυρίας μετά από αντιρρήσεις των ΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει οπωσδήποτε να υπάρξει εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία. Αλλά και η Ιαπωνία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Άρα έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη φαλαινοθυρία. Α ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ. Να πιέσουμε την Ιαπωνία να σταματήσει αυτή η άσκοπη και πεπαλαιωμένη παράδοση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριο Γουαλέντσα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να το συνδέσουμε με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεών μας με την Ιαπωνία για αυτή τη Συμφωνία Ελευθεροεμπορίου. Και γιατί. Και οι δύο πλευρές θέλουν να καταλήξουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Εντάξει. Αυτό το λέγαμε και πέρυσι και πρόπερσι, αλλά εμπάσπερτο. Η συμφωνία αυτή δεν είναι μόνο εμπορική όμω. Αν δούμε τι κάνει ο Τραμπ, που αποφάσισε να καταργήσει την συμφωνία TPP, χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία για να προωθήσουμε το στόχο γενικά συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Αν έχουμε καταλήξει όλα τα άλλα θέματα μέχρι το τέλο του χρόνου. Τι θα γίνει με αυτήν την αναφορά. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τι φάλαινε. Πρέπει να καταδικάσουμε εκπεφρασμένα όλες αυτές τις ε, δραστηριότητε φαλαινοθυρία. Αλλά μήπω θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ασκούμε επίση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των σχέσεών μα με την Ιαπωνία γενικά. Ο συνδυασμό και η ένταξη του θέματο αυτού στην ε, διαπραγμάτευση για την Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου δεν έχει καμία έννοια. Ιδιαίτερα αν πρόκειται να καταλήξουμε τον επόμενο μήνα σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες, τον, την οργάνωση αυτή για την προστασία των φαλενών και των δελφινιών. Είναι πολύ επίγον θέμα. Το 1982, όπως ξέρετε, η Διεθνής Επιτροπή Φάλαινο Θηρίας αποφάσισε να υπάρξει διακοπή όλων των δραστηριοτήτων φαλαινοθυρίας και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η απαγόρευση για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό αυτών και για να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Αλλά παρόλα αυτά η εμπορική φαλαινοθυρία συνεχίζεται από ορισμένες χώρες μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία. Και από τότε που εισήχθη αυτή η απαγόρευση η Ιαπωνία έχει δολοφονήσει πάνω από 20.000 φάλαινες και τα επόμενα 12 χρόνια θέλουν να σκοτώσουν άλλες 4.000. Πριν από 1,5 χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικά, κάλεσε την Ιαπωνία να σταματήσει να σκοτώνει οι φάλαινες. Και ενώ ήδη διαπραγματευόμασταν την Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου με την Ιαπωνία, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει κάθε διμερή και πολυμερή δυνατότητα για να ασκεί πίεση από τις Ιαπωνίας να σταματήσει και η Ιαπωνία συνεχίζει. Πριν από λίγες ώρες η οργάνωση Sea Shepherd ε, έβαλε στο ε, διαδίκτυο ένα φιλμ ε, που είναι πραγματικά απέσιο. Δείχνουν πώς σκοτώνουν με καμάκια φάλαινες. Και αυτό το φιλμ είχε γυριστεί πριν από πέντε χρόνια αλλά η αυστραλινή κυβέρνηση απαγόρευσε τη δημοσίευσή του γιατί θα ε, έβλαπτε τις σχέσεις της Αυστραλίας με την Ιαπωνία. Αυτά είναι άθλια. Η ελευθερία έκφραση και η προστασία, έκφρασης και η προστασία των ζώων είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι πιο σημαντικά από το βραχυπρόθεσμο οικονομικό συμφέρον κάποιων κυβερνήσεων. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τις εξηγήσει, για τη στήριξή τους. Και έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, μας εξηγήσατε πώς ε, τίθεται το θέμα αυτό στα πλαίσια των συναντήσεων για το ΣΥΤΕΣ και της ε, Επιτροπής ε, για την Φαλαινοθυρία. Αλλά πώς προσπαθείτε να πιέσετε στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων την Ιαπωνία, γιατί το Κοινοβούλιο αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία με την Ιαπωνία στο ψήφισμά του. Γιατί λοιπόν η Επιτροπή δεν βάζει κάποια ρήτρα για τη φαλαινοθυρία σε αυτή τη συμφωνία. Κάτι είπατε. Γιατί να μην πούμε ότι η Ιαπωνία και η Ένωση δεσμεύονται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους εντός των πολυμερών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Γιατί να αναφέρουμε την ε, φαλαινοθυρία αφού παραβιάζει και το ΣΥΤΕΣ και την ε, Συμφωνία για τη Φαλαινοθυρία η, η πρόεδρος. Ε, κοιτάξτε, η Κομισιόν περιέγραψε την άποψή της. Μπορεί να διαφωνείτε μαζί της. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση. Η Επιτροπή έφερε σαφώς την άποψή της. Ίσως διμερώς αν θέλετε μπορείτε να το συζητήσετε περαιτέρω. Δεν έχει έννοια να τους ζητήσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να έχουν και δύο διάθεση να αλλάξουν άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα της παράνομης φαλενοθυρίας, τόσο από πλευράς Ιαπωνίας όσο και από πλευράς Νορβηγίας έχει συζητηθεί α, ε, ορισμένες φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω λάβει το λόγο και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και φυσικά έχει περάσει και ψήφισμα κατά της Ιαπωνίας διότι παραβιάζει το παγκόσμιο μορατόριο για φαλενοθυρία. Έχει σφαγιάσει κυριολεκτικά πάνω από 20.000 φάλαινες προγραμματίζει να σφαγιάσει πάνω από 4.000 φάλαινες στο επόμενο διάστημα. Στην ουσία η Ιαπωνία κάνει ό,τι της γουστάρει. Δεν δίνει αναφορά σε κανέναν, θεωρεί ότι είναι υπεράνω του διεθνούς δικαίου και στο τέλος αποδεικνύεται ότι επειδή δεν λαμβάνονται μέτρα εναντίον της, ότι μπορεί να συνεχίσει να το κάνει και θα γίνει και χειρότερη και θα παραβιάσει και άλλες συμφωνίες. Εγώ ήθελα να συγχαρώ τον αναφέροντα διότι επιτέλους υπάρχει και κάποιος πολίτης ή μια οργάνωση πολιτών που έχει μαζέψει 267.000 υπογραφές και διαμαρτύρεται και φέρνει το θέμα εδώ. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον. Είναι ότι στο αίτημα της αναφοράς είναι στην ουσία να μπλοκάρει μια διεθνή συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας εάν δεν τεθεί το θέμα αυτό με αποφασιστικότητα. Δηλαδή, μέσα από το δικαίωμα της αναφοράς ο πολίτης είναι παρόν και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συνθήκες. Και μέσω της Επιτροπής Αναφορών μπορεί πλέον να ακουστεί η φωνή του και να μην έχουμε αποφάσεις για διεθνείς συμβάσεις πίσω από κλειστέ πόρτες. Πολύ δε περισσότερο σε ένα τέτοιο θέμα. Σημαντικό. Έχουμε δει τις σκηνές οι οποίες διαδραματίζονται με τα καμάκια, πώς βάζουν τις φάλαινες, τι γίνεται. Απέσια πράγματα δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη εποχή να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτή η διαδικασία. Και έχουν βρει και ένα άλλο κόλπο τώρα. Λένε ότι μπορεί να κάνουν δίθεν ε, φαλαινοθυρία για επιστημονικούς σκοπούς. Αυτό είναι ένα άλλο παραμύθι το οποίο έχουν στήσει τώρα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και αυτό ισχύει και για την Ορβηγία Και να πω στην Κομισιόν ότι το κρέας από φάλαινες που σφάζουν στην Ορβηγία περνάει μέσα από λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μου κάνει εντύπωση πώς περνάει από αυτά τα λιμάνια. Κατά παραβίαση της οδηγίας που υπάρχει. Και ποιος εμπλέκεται. Λοιπόν, ξεκάθαρα το μήνυμα από πλευράς μας είναι ότι πρέπει να πάρει ένα μήνυμα η Ιαπωνία. Και για να πάρει μήνυμα πρακτικό πρέπει να υπάρχουν πρακτικά αποτελέσματα. Και για να υπάρξουν πρακτικά αποτελέσματα πρέπει να μπει στην κουβέντα για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωση Ιαπωνίας. Μόνο έτσι θα καταλάβουν. Βεβαίω υπάρχουν επιχειρήματα ότι αυτή είναι μια σημαντική συμφωνία η οποία πρέπει να προχωρήσει. Ναι, δεν μπορεί όμως η ανθρωπότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείνει τα μάτια στη σφαγή των φαλενών και για λόγους οικολογικούς και για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και για λόγους τάξεως. Επομένως εγώ υποστηρίζω την αναφορά, επιμένω ότι πρέπει η Επιτροπή να βρει τρόπους να το θέσει το θέμα και να εξηγήσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα. Αν, και τελειώνω, σε αυτή τη συνεδρίαση κλείσουμε αυτή την αναφορά εγώ σας λέω ότι θα αποθρασινθεί η Ιαπωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα αποθρασινθεί και η Νορβηγία. Για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να στείλουμε μήνυμα αποφασιστικό. Τουλάχιστον όσον αφορά τη δικιά μου πλευρά, εγώ υποστηρίζω την αναφορά αυτή η οποία πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, να κρατηθεί ανοιχτή και να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει ακόμη πιο δραστήρια, πιο creative, πιο imaginatory, να βρει τρόπους να θέσει τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Now... Ε, και τώρα η Άγχελα. Και μετά πρέπει να κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Σε παρακαλώ, Άγγελα. Θα είμαι πολύ σύντομη. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μαριά. Και διαφωνώ πλήρω με τον κύριο Βαλέντσα. Γιατί τι αξιοπιστία μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν σε μια εμπορική συμφωνία, μέσω μια εμπορική συμφωνία. επιστρέψει επιτρέπουμε την εξαφάνιση ενό είδου ή όλε αυτέ τι βαρβαρότητε που γίνονται. Δίνουμε την εντύπωση ε, ότι δεν ακούμε του πολίτε που μα λένε όχι. Ε, και το μόνο που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τα, συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα ε, συγκεκριμένων παικτών. Ε, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τέτοια εικόνα εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι έχουμε 250.000 υπογραφέ που λένε αυτό που λένε και θέλουν να θέσουμε συγκεκριμένου όρου σε αυτή την ε, συνθήκη. Ε, θα χάσουμε και το κύριο που έχουμε σε τρίτες χώρες αν επιτρέπουμε ε, να, τέτοιες συνεχείς και επανειλημμένες παραβάσεις ε, των διεθνών κανόνων και της διεθνούς νομοθεσίας. Οπότε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Okay, fine. Let, let... Ωραία κύριε Φέντερ, έχετε ξανά το λόγο. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, πολύ σύντομα όμως παρακαλώ. Ορισμένα τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ πολύ την ε, Κομισιόν για την θέση της ε, σε συνόδους της ε, ΣΥΤΕΣ σε ό,τι αφορά την Ιαπωνία. Μα ικανοποιεί η δουλειά που έχει γίνει ω τώρα, αλλά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν παραπάνω. Ε, το θέμα θα πρέπει να θυγεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της ελεύθερης ε, συμφωνίας ελευθερομπορίου. Ε, είπατε ότι χρειάζεται, ε, χρειάζονται ε, δύο για να χορέψεις ε, το τάγκο, αλλά αν δεν ρωτήσει τον άλλον αν θέλει να χορέψει, δεν θα ξέρεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρος κάτι ανορθόδοξο. Ο τρόπος που ε, η επιλογή θα πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι πολιτική. Η Κομισιόν έκανε ό,τι μπορεί και έχω πλέον δύο διαφορετικές ε, θέσεις στην Επιτροπή μου. Να σας προτείνω το εξής, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να στείλουμε μια πολιτική επιστολή στον Επίτροπο. στην Επιτροπή, στην κυρία Μάλστρομ. Να της πούμε ότι συζητήσαμε το θέμα σήμερα και ότι ανησυχούμε πολύ. Ασφαλώς και θέλουμε να προχωρήσουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά ότι θέλουμε να πάρει και αυτό το θέμα υπόψη, ότι είναι ανησυχία 268.000 πολιτών στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να παραχώσει ένα σιρτάρι και να το ξεχάσει. Αυτή είναι η πρότασή μου και βλέπω ότι πολλοί συμφωνούν. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι πρέπει στην επιστολή στην Κομισιόν να αναφερθούμε και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει μια σαφήνεια για το θέμα αυτό και από εκεί και πέρα να ζητήσουμε την μέγιστη εφαρμογή του ψηφίσματος σε σχέση και με την πρόταση που έχουμε εδώ από την αναφορά. Και αυτό να είναι το μήνυμα, το πνεύμα, το πολιτικό πνεύμα, όπως είπατε, προς την Κομισιόν. Από εκεί και πέρα ε, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να στείλουμε την αναφορά μας και για περισσότερη διαδικασία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Νομίζω ότι αυτά θα είναι αρκετά. Ε, Ωραία. Αυτό είναι μπορούμε να κάνουμε και ο αναφέρον φαντάζομαι θα ικανοποιηθεί από αυτό. Είναι, συνήθως δεν κάνουμε τέτοιου είδους πράγματα. Ε, μιλώ για μια προσωπική επιστολή προς την Επίτροπο. Συνήθως αυτό που στέλνουμε είναι ε, όργανο προς όργανο. Ε, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε, που υπογραμμίσατε τη σημασία του θέματος. Περνάμε στο σημείο 11. Παρουσίαση της μελέτης, παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, εργαλεία και προκλήσεις. Καλώς ορίζω την εκπρόσωπο την κυρία Μπαγεστέρος. Νομική και πολιτική σύμβουλο. Παρακαλώ. Um, Καλημέρα σας. Μάρτα Μπαγιεστέρος ονομάζομαι, είμαι δικηγόρος και σύμβουλος στην Μιλιέ, μια εταιρεία η οποία εργάζεται στα πλαίσια της παρακολούθησης, της εφαρμογής και της επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας σε πάρα πολλές πτυχές, αλλά κυρίως στον περιβαλλοντικό τομέα. Συνεργάζομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πάνω από 8 χρόνια, σχεδόν σε αιτήσια μάλιστα βάση, εξετάζω την αιτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθώ να προχωρήσω σε μία αξιολόγηση του πώς έχει η κατάσταση και κατά αυτόν τον τρόπο έχω μια ξεκάθαρη ιδέα για τα βασικότερα σημεία της εξέλιξης της επιβολής της κοινωνικής νομοθεσίας, επί την οποία θα ήθελα να επικεντρωθώ βέβαια σήμερα, στη σημερινή μου παρουσίαση. Θα αναφερθώ λοιπόν καταρχάς στους βασικούς παράγοντες που έχουμε, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε δει σε σχέση με τη δική του την εμπλοκή στην εφαρμογή και επιβολή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια θα ήθελα να διατρέξω τα σημαντικότερα σημεία που έχουν να κάνουν με την επιβολή, τη μεταφορά, την, τα μέσα υποστήριξης μεταφοράς, καθώς επίσης και την πολιτική επιβολή. Λοιπόν, εν ίδια αρχής, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το κράτος δικαίου. όπου λέγεται ότι η διασφάλιση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά του κράτους δικαίου, γιατί έχει να κάνει με τις καταστάσεις εκείνες όπου οι δημόσιες αρχές πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια των νόμων, σεβόμενες τις αξίες της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτό συνδέεται με τις έννοιες της νομιμότητας, ασφάλειας δικαίου, της απαγόρευσης αυθαίρετων αποφάσεων και θεωρώ ότι οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για κάποια από τα επιχειρήματα τα οποία θα σας παραθέσω λίγο αργότερα. Η σημασία της εφαρμογής, της διασφάλισης εφαρμογής της κοινωτική νομοθεσίας σε κάθε κράτος μέλος ουσιαστικά βασίζεται στους ίδιους τους στόχους της κοινωτική νομοθεσίας η διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας διασφαλίζει τελικά ότι οι στόχοι αυτή πολιτικής όντως επιτυγχάνονται στην πράξη. Και κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε να έχουμε αρνητικό αντίκτυπο, δηλαδή αποφεύγεται τελικά ο αρνητικός αυτός αντίκτυπος που είναι και ο λόγος έγκρισης τελικά της ίδιας νομοθεσίας. Επίσης, εφόσον αναφερόμαστε στο κοινοτικό δίκαιο, στο ενωσιακό δίκαιο, δηλαδή αναφερόμαστε στην νομοθεσία που εγκρίνεται και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα τελικά και αν έχουμε ένα, δύο και περισσότερα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν νομοθεσία κατά τον ίδιο τρόπο με τα υπόλοιπα μέλη, τότε αυτό από μόνο του μπορεί να ταράξει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και ένας ακόμα σημαντικός λόγος είναι η ίδια η εξοπιστία της Ένωσης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει μια κάποια νομοθεσία, τότε η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται. Η Ένωση πρέπει να έχει τα μέσα για να επιβάλλει αυτή τη νομοθεσία εν συνεχεία. Ποιος είναι υπεύθυνο λοιπόν για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Έχουμε τρία θεσμικά όργανα με μια διοργανική συμφωνία, Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο, που θεωρούν ότι πλέον έχουν κοινή ευθύνη για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό το έχει τονίσει και το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση 1999 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ιταλίας. Πώς έχει λοιπόν τώρα η κατάσταση σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, σύμφωνα πάντα με τις συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με συγκεκριμένους τομείς όπως με το τομέα του περιβάλλοντος. Τώρα τα κράτη-μέλη εμπλέκονται προφανώς στην νομοθετική διαδικασία, εγκρίνουν και αυτά ενωσιακή νομοθεσία. Το Συμβούλιο, όπως ξέρετε, είναι συνομοθέτης μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η νομοθεσία επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες στα κράτη-μέλη. Το ίδιο το Συμβούλιο έχει διαπραγματευτεί για πάρα πολλά χρόνια για την νομοθεσία αυτή και φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του. Βέβαια, τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε καταδεικνύουν ότι πολλές φορές η εφαρμογή της νομοθεσίας παραμένει σημαντική πρόκληση. Έχουμε περίπου 840 νέες υποθέσεις που αφορούν τη μεταφορά νομοθεσίας, μη σωστή, μη ορθή μεταφορά νομοθεσίας και έχουμε περίπου 800 νέες διαδικασίες U-Pilot και περίπου 980 νέες διαδικασίες επί παραβάση. Και αυτά κάθε χρόνο. Τα αριθμητικά αυτά δεδομένα δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν εφαρμόζουν τελικά την κοινοτική νομοθεσία. Θα μπορούσαμε να δούμε και κάποια περαιτέρω αριθμητικά δεδομένα, ποια είναι η γενικότερη τάση το 2015 και το 2016 βλέπουμε ότι ο υψηλότερος αριθμός διαδικασιών επί παραβάση και διαδικασιών EU Pilot είχε να κάνει με το τομέα του περιβάλλοντος, αλλά και με το τομέα των μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς, αλλά κυρίως με το τομέα του περιβάλλοντος. Αν πάρουμε λοιπόν το τομέα του περιβάλλοντος, τα βασικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν εκεί το 2015 για τα EU Pilot ήταν η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση των υδάτων και η φύση. Το 2016 ήταν πάλι τα ύδατα, η προστασία της φύσης και οι χημικές ουσίες. Το 2015 είχαμε 120 διαδικασίες παραβάση για περιβαλλοντικά θέματα, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, τα ύδατα και τις χημικές ουσίες, ενώ είχαμε περίπου 90 τέτοιες περιπτώσεις το 2016. Οι δράσεις που αναλαμβάνει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκούν ή ε, μήπως είναι τελικά απλώς η κορφή του παγόβουνου. Αν διαβάσουμε άλλες εκθέσεις, όταν διαβάζουμε άλλες εκθέσεις, για παράδειγμα για την Ελλάδα, όπου έχουμε συστηματικές καταγγελίες από μη κυβερνητικέ οργανώσεις όπως η WWF αλλά και από μονομένους πολίτες οι οποίοι αναφέρονται σε εκθέσεις εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια συστηματική τάση έγκρισης αποφάσεων για την ε, αποστεριώρη νομοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων. Κτίσματα λοιπόν τα οποία ήταν αυθαίρετα, παράνομα. Και αυτό βέβαια αντιβαίνει και στο κοινοτικό δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο. Βέβαια βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει καμία δράση στη συνέχεια, ενδεχομένω να μην έχει του πόρου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλύψει όλε αυτέ τι περιπτώσει παράβαση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπουμε ότι εν προκειμένου η παράβαση αυτή έχει πλέον συστηματικό χαρακτήρα. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και ήδη από το 2000 το έχει θέσει αυτό προτεραιότητά της. Στην ανακοίνωσή της για τη διακυβέρνηση του 2002, 7, 8 και 10 αναφέρεται ότι η διασφάλιση της εφαρμογής της νοσιακής νομοθεσίας αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, είχαμε κάποιες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους, τρίτους, ένας από τους τρεις με στόχους για την εφαρμογή της νοσιακής ομοθεσίας μειώνει τελικά τη χρήση της διαδικασίας επί παραβάση. Στη νέα ανακοίνωση που γίνεται για την πολιτική για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου το 2015 αλλά και το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς προτεραιότητας. Η ανάληψη δράσης πρώτον, παρακολούθηση της εφαρμογής της νοσιακής νομοθεσίας, δεύτερον, επίλυση προβλημάτων προκύπτουν με τα κράτη-μέλη και τρίτον, ανάληψη. Η κίνηση μάλλον διαδικασία σε παραβάσεις, αυτό κρίνεται αναγκαίο. Αν δούμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2016, λέγεται ότι θα αναλυφθεί δράση όταν πραγματικά αυτό μπορεί να αποφέρει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Όταν υπάρχει μία πολιτική προτεραιότητα όταν πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη. Ενδεχομένω θα μπορούσε λοιπόν να αναλάβει μια τέτοια δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα προκειμένου. Επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι θα ξεκινήσει διαδικασίε επιπαραβάσει στο μέλλον χωρίς να περνάνε από τη διαδικασία EU Pilot και λέει επίσης ότι θα βασίζεται στο εργαλείο αυτό, στο μηχανισμό EU Pilot, όταν αυτός ο μηχανισμός κρίνεται χρήσιμος για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μία σημαντική αλλαγή πλέον στην πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πρέπει να το γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια λοιπόν τώρα της στρατηγικής αυτής που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τελευταίες της αυτές ανακοινώσεις υπάρχουν και κάποια επιπλέον στοιχεία, κάποιες επιπλέον πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε μια μελέτη όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας επιβολής για τον τομέα του περιβάλλοντος. Εκεί πέρα για παράδειγμα βλέπουμε ότι ε, η πολιτική επιβολή νομοθεσίας θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξοικονομήσουμε τεράστια ποσά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποδεικνύεται επίσης ε, στα πλαίσια της επισκόπης εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τελικά για ποιους λόγους τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την ουσιακή νομοθεσία, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος που είναι τόσο προβληματικός. Το ενδιαφέρον εδώ είναι να δούμε σε σχέση με τους προφανείς λόγους, όπως για παράδειγμα έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων, έλλειψη διοικητικής ικανότητας, έλλειψη χρηματοδότησης. Πέρα από τους προφανείς αυτούς λόγους πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα συστήματα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν είναι διαρθρωτικό δεν είναι ότι μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει απαραίτητη βούληση από ένα κράτο μέλο για να επιβάλλει την νομοθεσία και ενδεχομένω να υπάρχει μια βελτίωση. Αν δεν υπάρχουν συστήματα για τη διασφάλιση μόρφωση, το πρόβλημα γίνεται αυτόματα διαρθρωτικό και επομένω δεν πρόκειται ποτέ να επιβάλλεται σωστά η νομοθεσία. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν και απαραίτητε κυρώσει για να διασφαλίσει την εφαρμογή τη νομοθεσία. Ένα ακόμα λόγος που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ε, πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό μέσω της βελτίωσης του νομοθετικού έργου. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την στρατηγική αυτή Better Regulation για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, όπου κάθε νομοθεσία εγκρίνεται τελικά μόνο αφού γίνει πρώτα αξιολόγηση αντικτύπου και έπειτα είχαμε και την διαδικασία REFIT, για την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα δηλαδή της κοινοτικής νομοθεσίας και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε νέες πλατφόρμες για να έχει ε, μια καλύτερη συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τεχνική αυτή πλατφόρμα συνεργασίας στον τομέα του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει κατά αυτόν τον τρόπο τις αιτησεις εκθέσεις και ξεκινά όπου το κρίνει αναγκαίο τις ε, διαδικασίες παραβάση ή χρησιμοποιεί και το μηχανισμό EU Pilot, ο οποίος θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζωτικό ρόλο γιατί έχει αρμοδιότητες ελέγχου έναντι της Επιτροπής αλλά και ως νομοθέτης να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας λαμβάνει χώρα και έχει διάφορες δυνατότητες. Ορισμένες θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμες. Για παράδειγμα, Το γεγονό ότι επανεκλέγεται κάθε πέντε χρόνια ε, είναι βασικό για την δημοκρατική του νομιμοποίηση. Βέβαια αυτό δεν βοηθάει ορισμένε φορέ στη συνέχιση τη παρακολούθηση των θεμάτων. Αλλά έχουν πολλέ πηγέ πληροφοριών, μελέτε που εκπονούνται συνεχώς. Έχουν τα τμήματα πολιτικής που εκπονούν εκθέσεις Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ε, συνεχή πληροφόρηση για την εξέλιξη της κατάστασης. Αυτό νομίζω βοηθάει πολύ. Βοηθάει και την Επιτροπή. Και το Κοινοβούλιο. Και βοηθάει επίσης και το ότι έχει άλλες δυνατότητες όπως τις εκθέσεις πρωτοβουλίας που είναι πολύ χρήσιμες αλλά ορισμένε φορές υπολείπονται των εξελίξεων. Ίσως θα μπορούσε το Κοινοβούλιο να μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικό μέσω εκπόνησης ταχύτερα εκθέσεων πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, υπάρχει μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη. ενώ ε, εμείς έχουμε περάσει τώρα στο refit. Αν είχε γίνει νωρίτερα αυτή η έκθεση θα είχε βοηθήσει περισσότερο. Άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο. Παρακολουθεί την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προφανώς, αλλά επειδή εκπροσωπεί τους πολίτες, λαμβάνει και τις αναφορές από τους πολίτες. Πόσες αναφορές έχουν καταλήξει σε ανάληψη δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως βλέπετε, μειώνεται ο αριθμός τους. Νομίζω ότι ο ρόλος της Επιτροπής σας είναι ζωτική σημασίας. Αλλά θα μπορούσατε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητά σας εάν Παρακολουθείτε συνεχώς όλες τις αναφορές τις οποίες έχετε ε, αντιμετωπίσει απαιτώντας ε, να λαμβάνετε συνεχή πληροφόρηση, να εξελίσσετε κατάσταση και να ενημερώνετε και τον αναφέροντα για το τι συμβαίνει. Και οι πολίτες της Ένωσης είναι κρίσιμοι. Με βάση το άρθρο 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχική δημοκρατία είναι βασική αρχή της Ένωσης. Άρα, οι πολίτες παρακαλούνται να αποστέλουν πληροφόρηση για διάφορους τομείς που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, μεταξύ των οποίων είναι και η εφαρμογή του ενωσιακού νόμου. Φέτος, δηλαδή πέρυσι, αυξήθηκε ο αριθμός ε, των ε, ετοιμάτων και ενστάσεων που υπέβαλαν οι πολίτες ε, αυξάνεται συνεχώς από το 2011. Αλλά δεν είναι σαφές Τι επίπτωση είχαν αυτές οι 3.700 ενστάσεις. Η Επιτροπή τις θεωρεί θεμελιώδη πηγή πληροφόρησης, αλλά τονίζει ότι πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ποιος είναι ο στόχος της διαδικασίας επί παραβάση. Ε, πρέπει να αφορά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. Αυτό ίσως θα μπορούσε να το αμφισβητήσει το Κοινοβούλιο. Γιατί η διαδικασία επί παραβάση πρέπει να αφορά μόνο ευρύτερα θέματα. Γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν ένα μέσο για να αντιμετωπίζονται όλες οι παραβιάσεις περιβαλλοντικού δικαίου. Γιατί και τι σημαίνει ε, θέματα ευρύτερης σημασίας, ε, πώς θερμινεύει η Επιτροπή, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Γιατί ποια είναι η κατάσταση των πολιτών που υποβάλλουν παράπονα. Στη, δεκαετία του 80 και του 90 ο διάλογος ε, με τους ε, υποβάλλοντες ενστάσεις ήταν πολύ πιο στενός. Ήμουν παρούσα και το διαπίστωσα αυτό. Όταν υποβάλλεται ένα παράπονο, μια ένσταση, η Κομισιόν ζητούσε περισσότερη πληροφόρηση ή και συζητούσε τα επιχειρήματα του πολίτη για να μπορέσει να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλαν τα κράτη-μέλη. Αλλά τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες. Ο πολίτης που υποβάλλει παράπονο δεν λαμβάνει καμία ενημέρωση. Πέραν ε, της ε, ενημέρωσης ότι ελήφθη η ένσταση ενώ θα έπρεπε σε κάθε διαδικαστικό βήμα να ενημερώνει τον πολίτη. Δεν συμβαίνει πάντα, θα έπρεπε να συμβαίνει. Και κατά την περίοδο εξέτασης μέχρι να ληφθεί απόφαση να κλείσει το θέμα ή να σταλεί επίσημη επιστολή προειδοποίησης, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το έτος. από τις 3.700 ε, ε, διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2016 μόνο 270 οδήγησαν σε ενωσιακά πιλωτικά προγράμματα. Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται ότι 3.026 έκλεισαν. Αλλά ίσως να μην ήταν ε, αναφορές του 2016. Λοιπόν, από 3.783 ενστάσεις, μόνο 270 κατέληξαν σε κάποια δράση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πολλές από τις ενστάσεις αφορούσαν θέματα που δεν ήταν ενωσιακής αρμοδιότητας ή αρμοδιότητας της Επιτροπής ή δεν ε, ενέπιπταν στην ε, ενωσιακή νομοθεσία. Που φαίνονται πολύ ψηλά αυτά τα νούμερα, αλλά δεν αναφέρεται αναλυτική πληροφόρηση στην έκθεση. Ίσως θα χρειαζόταν λοιπόν περισσότερη πληροφόρηση. Το Κοινοβούλιο, σε ένα ψήφισμά του, καλεί να εγκριθεί κανονισμός που να καθορίζει τους κανόνες για τις προσφυγές επί παραβάση αλλά θα μπορούσε να ζητήσει και περισσότερη πληροφόρηση στην επόμενη έκθεση της Επιτροπής. Η τάση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είναι πτωτική. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται η μη μεταφορά ή η καθυστερημένη μεταφορά. Είχαμε 790 τέτοιες περιπτώσεις. Να αναφερθώ στα κύρια θέματα. η Κομισιόν δεν εξετάζει μόνο πόσο χρόνο παίρνει η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αλλά εξετάζει αν γίνεται και σωστά η μεταφορά. για να το κάνει αυτό έχει μελέτες ε, συμμόρφωσης και πίνακες συσχέτισης. Αυτό θα έπρεπε να είναι ευθύνη των κρατών μελών. Εκείνοι ενημερώνουν την Κομισιόν για, για τα νομοθετήματα μεταφοράς. Πιο εύκολα λοιπόν θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν ποιο άρθρο μεταφέρει ποια ρήτρα της οδηγίας. Στην πραγματικότητα όμως το Συμβούλιο ποτέ δεν δέχτηκε να επιβληθεί υποχρέωση στα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι τέτοιο. Ναι, μένει, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο το έχουν ζητήσει, αλλά δεν έχει γίνει. Και τελικά τις μελέτες αυτές τις κάνει η Επιτροπή για να εξετάσει πώς γίνεται η μεταφορά των ενωσιακών νομοθετημάτων. Αλλά αυτές οι μελέτες δεν δημοσιοποιούνται, θεωρούνται εμπιστευτικέ. Γιατί είναι πολύ χρήσιμες για ενδεχόμενε προσφυγές. Από την άλλη μεριά βέβαια είναι δημόσια έγγραφα, οπότε μπορούν να γίνουν αιτήματα πρόσβασης. Είναι αναλύσεις της ε, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή όχι αυτές τις μελέτες. Τις κάνουν κυρίως εταιρείε συμβούλων. Άρα δεν ε, είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν μετά ούτε να συμφωνήσει με τα απορίσματά τους, ούτε να τις εφαρμόσει. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Κομισιόν έχει επαρκείς πόρους για να μπορεί να κάνει αυτές τις μελέτες μέχρι να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη να τις κάνουν τα ίδια και θα μπορούσε να πιέσει την Κομισιόν να τις δημοσιοποιεί για να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων μεταφοράς. Καταλήγοντας, να πω δύο λόγια για τη διαδικασία επί παραβάση. έχουν μειωθεί αυτές οι διαδικασίες. Αυτή η μείωση βέβαια κάπως ε, αντισταθμίστηκε πέρυσι. Αλλά είναι σαφές ότι η διαδικασία επί παραβάση είναι πολύ αποτελεσματική και έχει και αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Αλλά βέβαια δεν βασίζεται σε νομικά δεσμευτικούς κανόνες Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εμείνει ενώπιον της Επιτροπής για να υποβάλει πρόταση κανονισμού ούτως ώστε να υπάρξουν νομικά δεσμευτικοί κανόνες. Ευχαριστώ πολύ επιτρέψτε μου να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που μόλις είπατε. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, μειώνονται, λέτε. Αν ε, λάβετε υπόψη σας τις διαδικασίες παραβάση, ε, είμαστε σε διάλογο με την Κομισιόν. Η διαδικασία επί θα πρέπει να είναι όσο λιγότερες γίνεται. Αν, αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα νωρίτερα και χωρίς να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, καλύτερο. Γιατί θα πρέπει να ε, σέρνουμε τα κράτη-μέλη ε, στο δικαστήριο αν μπορούμε να ρυθμίσουμε αλλιώ τα προβλήματα. Αυτό είναι σε σελίδα 27. Η τελευταία παράγραφος πριν το 1, 2, 4 θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Συμφωνώ, διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ απόλυτα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή κάνουν πολλές ε, ε, πληροφοριακές ε, επισκέψεις, υποβάλλουμε μικρά ψηφίσματα, προφορικές ερωτήσεις, παρόλο ότι μπορεί να μην οδηγούνται, να μην οδηγούνται τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή Παραβάση. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να σχαροποιεί. Ο στον στην, Επίτροπο της στην εκπρόσωπο της Κομισιόν Ρενέ Σλότσες. Ε, Ο κύριος Ρενέ Σλότσες. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει κυρία Βαγεστέρο σε αυτή τη δουλειά. Ε, κάνει φανερή την πρόοδο που έχει συμβεί σε θέματα συμμόρφωσης. Ε, βέβαια εντοπίζει και, τα, και τις προκλήσεις η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσία είναι απαραίτητη προκειμένου οι ευρωπαϊκές πολιτικές να ε, δείξουν την αξία τους. Η σωστή εφαρμογή τη νομοθεσία εξασφαλίζει ότι ε, ε, και οι εταιρείε και τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να χαίρουν των δικαιωμάτων τους. Πρέπει λοιπόν να διατρήσουμε ως υψηλή προτεραιότητα της Κομισιόν την συμμόρφωση με το δίκαιο. Υπάρχουν πολλές σημαντικές εξελίξεις όμως μια πιο στρατηγική, για παράδειγμα, προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις ε, διαδικασίες παραβάση που ε, παρουσιάσαμε το 2016. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο απαντήσαμε σε πολλά θέματα που έχειρατε στη μελέτη σας. Η πολιτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου είναι πιο στρατηγική, εστιάζεται στις ε, πιο σημαντικές παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των πολιτών. Εκεί δηλαδή μπορούμε να δούμε τη διαφορά. Ε, όταν η παραβίαση ε, εμποδίζει τους βασικούς στόχους της ε, νομοθεσίας, εκεί δρούμε γρήγορα και αυστηρά. Ε, πώς ερευνούμε γρήγορα υποθέσεις μη σωστής μεταγραφής ή απουσίας μεταγραφής. Επίσης περιπτώσεις που τα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει συνέχεια στι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, ή πλήττονται συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, ε, όταν δεν εφαρμόζουν αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που έχουν εκφέρει γνώμη υπέρ της επικράτησης του κοινοτικού δικαίου πάνω από το εθνικό δίκαιο. Βέβαια, δεν μπορούμε να επιλύουμε όλα τα προβλήματα μέσω διαδικασιών προσφυγή, αυτό όμως ε, δεν σημαίνει ότι θα απογοητεύσουμε αυτούς που ε, έχουν καταγγείλει παραβάσεις. Πολλές ε, φορές όμως μπορούν να χρησιμοποιήσουμε άλλους πιο κατάλληλους μηχανισμούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις και μόνο όταν υφίσταται επαρκής νομική προστασία η Κομισιόν θα παραπέμψει τους καταγγέλλοντες σε, άλλους, σε άλλα όργανα και άλλα επίπεδα που είναι ε, πιο κατάλληλα. Όπως σας είπα, ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την συνεισφορά των πολιτών και των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των παραβιάσεων, όμως ε, ε, θα πρέπει να τήρουμε το μέτρο. Πολλοί υποβάλλουν καταγγελίες και ελπίζουν ότι θα λάβουν οικονομική αποζημίωση. Όμως ο βασικός ε, λόγος μιας διαδικασίας που παραβάσει δεν είναι η αποζημίωση σε συγκεκριμένους μονομενούς πολίτες, αλλά το να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπως σας είπα όμως θα εξακολουθήσουμε να χειριζόμαστε περιπτώσεις ε, μεμονωμένων πολιτών που ε, κρύβουν ή υποδεικνύουν γενικευμένες πρακτικές ε, παραβίασης, ε, όπως επίσης και στην περίπτωση που δεν υφίστανται άλλοι καλύτεροι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Οπότε η ιδέα είναι ότι ορισμένα μεμονωμένα ζητήματα θα παραπέμπονται σε πιο τοπικό επίπεδο, ενώ πιο συστημικά ζητήματα, πιο γενικευμένη σημασία ζητήματα θα τα χειριζόμαστε εμείς μέσω διαδικασιών επί παραβάση. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα προσιλωμένοι για την ε, προάσπιση των προτύπων ε, διοικητικής συμπεριφοράς ε, και οποτεδήποτε υπάρχουν καταγγελίες σε εθνικό πεδίο για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες ε, ε, διαδικασίες καλής διοίκησης, χρηστής διοίκησης. Τώρα πια επίσης οτιδήποτε, ανα, για οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνουμε κατόπιν καταγγελίες θα ενημερώνουμε τον αναφέροντα χωρίς να μας το ζητήσει. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε να μην ακρηγορήσω. Υπίσταται ένα πλαίσιο για την προστασία των καταγγελόντων στην ε, διαδικασία παραβάση σε συνδυασμό με τον κώδικα καλής δικητικής ε, ε, συμπεριφοράς τον οποίο είμαστε δεσμευμένοι. Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι τα συμφέροντα όλων μπορούν να την υπόψη από εμά. Έχουμε λοιπόν οριζόντιους κανόνες που διέπουν τη δική μας διοικητική συμπεριφορά. Οπότε δεν θεωρούμε ότι ένα οποιοδήποτε άλλο νομοθετικό κείμενο ε, που θα κωδικοποιεί την, ε, το διοικητικό νόμο, τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες θα ήταν χρήσιμο. Μήπως έχετε τελειώσει να κλάβω έτσι με αυτόν τον τρόπο την σιωπή σα, Γιατί δεν θα έχουμε διερμηνία σε λίγο και έχουμε άλλο ένα μέλος που θέλει το λόγο. Γι' αυτό ε, ε, περνούσε εντάχει ε, πολλά από τα θέματα. Έχουμε πολιτικές που θα ενισχύσουν το καθεστώς οικονομικών κυρώσεων προκειμένου να αυτό να αποτελέσει κίνητρο για γρηγορότερη ψημόρφωση εκ μέρους των κρατών μελών. έχουμε προσαρμόσει τις διαδικασίες μας για τη διαδικασία EU Pilot. Η χρήση θα γίνει πιο διαρθρωμένη. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Οπότε, ευχαριστούμε για τη μελέτη. Έχουμε ορισμένα ζητήματα σε σχέση με κάποια από τα πορίσματα. Για παράδειγμα, ο αριθμός των ε, αναφορών ε, που οδήγησαν αυτές τις διαδικασίες παραβάση. Εμείς αναφέρουμε επτά παραδείγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο επτά αναφορές που οδήγησαν σε διαδικασίες παραβάση. Ήταν επτά παραδείγματα. Ε, επίσης λέτε ότι διασυνδιαλεγόμαστε με τους καταγγέλλοντες ή όταν κλείνουμε μια υπόθεση δεν ε, δίνουμε την αιτιολογία. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό, ότι ισχύει αυτό. Ε, θα το δείτε στην έκθεση του 2016 ότι αναφέρουμε τους λόγους και ε, πριν κλείσουμε οποιαδήποτε υπόθεση, έτσι κι αλλιώς αναφέρουμε τους λόγους μας στον καταγγέλλοντα και του δίνουμε την ευκαιρία να μας αντικρούσει. Έχουμε δύο θέματα σε σχέση με τη μελέτη που η θέση μας διαφέρει ζητάτε να ε, παρακολουθούμε καλύτερα την εφαρμογή του, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι, μας, ε, ο, μας ελέγχει, καθώς επίσης ελεγχόμαστε και από το ελεγκτικό συνέδριο. Όμως η διαδικασία επί παραβάση έχει μια διμερή φύση ε, μεταξύ της Κομισιόν και του κράτους μέλους. Οπότε ε, υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια Το ίδιο ισχύει και για την διαδικασία EU Pilot πρώτης ε, ε, ε, προσφυγή στην διαδικασία παραβάση. Χρειάζεται και εκεί να εξασφαλίζεται το απόρριτο. Παρ' όλα αυτά έχουμε λάβει για μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας. Το αναγνωρίζει και η μελέτη. Έχουμε ένα πολύ καλό site στο ίντερνετ με μια μηχανή αναζήτησης ε, για συγκεκριμένες περιπτώσεις και υποθέσεις διαδικασιών επί παραβάση. Οπότε ε, έχουμε πολύ συχνά διαδικασία επί παραβάση αποτελούν αντικείμενο ε, συνεντεύξεων τύπου. Οπότε πράγματι μεριμνούμε, μεριμνούμε έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε τη διαφάνεια και προς το Κοινοβούλιο και προς τους πολίτες μας. Ε, σε περιπτώσεις που ζητείτε πρόσβαση σε έγγραφα, αν η διαδικασία παραβάση είναι σε εξέλιξη, ε, καθυστερούμε συνήθως την αποκάλυψη των εγγράφων μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία παραβάση. Τελειώνοντας και συνοψίζοντας, Μοιραζόμαστε το ε, ενδιαφέρον σας για τη σωστή εφαρμογή του, της ε, κοινωνικής νομοθεσίας και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you. And I can also... Σας ευχαριστούμε. Να πω πάντως ότι ε, και εμεί χαιρόμαστε γιατί είχαμε μια βελτιωμένη και πιο ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορα ζητήματα για τα οποία βλέπουμε πλέον ότι δεν υφίσταται λόγος να κινηθεί διαδικασία επί παραβάση. Έτσι λοιπόν μπορώ να απαντήσω και εγώ στη μελέτη αυτή. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Uh, minutes or... Δύο λεπτά έχω στη θέση μου κυρία Πρόεδρε. Okay. Ε, καταρχάς είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη και προφανώς έπρεπε να έχουμε περισσότερο χρόνο οι ευρωβουλευτές για να τοποθετηθούμε κι εμείς. Εγώ θέλω να θέσω ένα θέμα προς την ε, εισηγήτρια που έχει φτιάξει τη μελέτη και βεβαίως και στην Κομισιόν. Και αυτό το θέμα είναι η παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ελληνική κυβέρνηση και την Κομισιόν με αφορμή αυτό που ονομάζουμε μνημόνιο, Memorandum of Understanding. Διότι αυτό επιβάλλεται από τους δανειστές το Eurogroup προκειμένου να εγκρίνει χρηματοδότηση του ESM ή των δανειστών προς την Ελλάδα επιβάλλει ένα Memorandum of Understanding το οποίο είναι πάρα πολύ αναλυτικό και επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα. Μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, διάλυση του κοινωνικού κράτους, διάλυση των ε, νοσοκομείων και όλα αυτά παραβιάζουν δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα, human rights, τα οποία καθορίζονται από την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δικαίωμα περιουσίας, όταν σου μειώσει τη σύνταξη κατά 30, 40, 50% είναι το δικαίωμα περιουσίας. Το δικαίωμα ε, το δικαίωμα να διαβιώνει κανείς αξιοπρεπώς, το δικαίωμά του στην περιουσία του, ε, επιβάλλονται ρυθμίσεις τώρα για κατασχέσεις fast track και χάνεις την περιουσία σου. Και γίνονται και ιδιωτικοποίησει. Έχω θέσει λοιπόν επανειλημμένο στο θέμα αυτό εδώ, λέγοντα ότι παραβιάζεται η νομοθεσία. Και η απάντηση που δίνει η Κομισιόν λέει η Κομισιόν δεν ξέρει τίποτε. Διότι το Memorandum of Understanding δεν είναι, λέει, κοινοτικό δίκαιο. Και έτσι δεν δεσμεύεται η Κομισιόν να προστατεύσει τα, την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, λέει η Κομισιόν, ότι ο νόμος ο ελληνικός που εφαρμόζει το Memorandum of Understanding, το μνημόνιο δηλαδή, δεν έχει σχέση με το κοινοτικό δίκαιο. Και έτσι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη όπου παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και κανείς δεν προστατεύει τους Έλληνες πολίτες. Έχουμε δεκάδες petitions που έχουν έρθει εδώ για το ζήτημα αυτό. Και απαντάει η Κομισιόν ότι δεν ξέρει τίποτε. Πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Θεωρούσα ότι θα είχα χρόνο να το αναπτύξω. <laughs> Δυστυχώ αυτό το σοβαρό θέμα δεν μα δίνει τη δυνατότητα να το συζητήσουμε αναλυτικά. Θέλω στη μελέτη σα λοιπόν στο μέλλον να δείτε αυτή την πλευρά αναλυτικά, να τη μελετήσετε και εμεί βεβαίω πάντοτε θα τη θέτουμε εδώ. Την έχουμε θέσει και στον κύριο Τίμερ μα, τη θέτουμε και στην Κομισιόν και επιμένουμε. I'm going to finish in 30 seconds, really. Ε, η Κομισιόν οφείλει να ελέγξει την παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωση Είναι μέλος τη Τρόικας και τι λέει στην Ελλάδα. Εάν δεν εφαρμόσεις το Memorandum of Understanding, το μνημόνιο, δεν θα πάρεις δάνειο, δεν θα πάρεις τα χρήματα. Άρα η Κομισιόν είναι ο οργανισμός που ελέγχει την εφαρμογή των εντολών των δανειστών. Πάβει να είναι ο Guardian, να είναι ο φύλακας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε άλλη φορά πιο αναλυτικά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Άλλη φορά πρέπει να μιλάμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Now, thank you very, very much for... Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή μας αυτή συνεδρίαση και θα σας δω στις 3.30 μαζί με τους ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Οι, βοηθήσει θα σας πούνε σε ποια αίθουσα. Νομίζω ότι είναι στο κτίριο PHS. Καλό μεσημέρι, καλή όρεξη. Θα σας δω σύντομα πάλι.